Κυρίες και κύριοι, καλημέρα, το διάλειμμα τελείωσε και ξαναξεκινάμε τη δουλειά μας. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που ήρθαν εν και σας παρακαλώ να έχουμε ησυχία στην αίθουσα. Σήμερα έχουμε τις περισσότερες ψηφοφορίες εφόσον όλη την ημέρα θα έχουμε ψηφοφορίες ιδίως όσον αφορά τη συνέχιση των των ψηφοφοριών για τον προπολογισμό του επομένου έτους αλλά για να μας ανοίξει η όρεξη ξεκινάμε με δύο ψηφοφορίες σε διαφορετικά θέματα για τα οποία είμαστε αρμόδιοι είτε για γνωμοδότηση είτε για να προτείνουμε μια απόφαση επί της ουσίας στην Ολομέλεια. Θα δώσω λοιπόν αμέσως το λόγο στην Μπάρμπαρα Ματέρα η οποία θα μας παρουσιάσει διάφορα θέματα όπου ζητείται η βοήθεια του ε, Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Θα ζητήσω λοιπόν στην εισηγήτρια να είναι όσο το δυνατόν πιο, γρήγο, πιο σύντομη και ελπίζω ότι έτσι δεν θα είναι δύσκολη η ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη παρότι σέβομαι και τους διεθνείς για να με παρακολουθούν. Ήθελα λοιπόν να παρουσιάσω τρεις διαφορετικές περιπτώσεις στους συναδέλφους όπου ζήθηκε η κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την παγκοσμιοποίηση. Δύο αιτήματα από τη Δανία και ένα τρίτο αίτημα από την Ισπανία, Γαλλικία. Τα δύο δανέζικα αιτήματα είναι η Τάμφος, το ένα, που ζητάει 8 εκατομμύρια 8,9 εκατομμύρια για 1010 εργαζόμενους. Είναι μια επιχείρηση που κατασκευάζει ηλεκτρικές συσκευές και η Λίνακ που ζητάει 139 139 εργαζόμενοι 1,2 εκατομμύρια ευρώ περίπου το αίτημα της Ισπανίας Γαλλικία. Εδώ μιλάμε για 500 εργαζόμενους, 82 επιχειρήσεις, κλωστοϊφαντουργία. Ποσό 1,85 εκατομμύρια ευρώ. Δίνοντας συνέχεια σε αιτήματα του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής ε, Προπολογισμών προς την Κομισιόν, η Κομισιόν ε, αναζήτησε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης σχετικά με, την, με τις με πληρωμές ως προς το Ταμείο. Στο 1α βρέθηκε η λύση για το πρόγραμμα καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας και για το πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που είπατε να βρεθεί τρόπος να δοθεί χρόνος για περισσότερη συζήτηση για το θέμα αυτό στο μέλλον. Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται για τις κινήσεις αυτές της Κομισιόν μου έστειλαν στοιχεία. Τρεις ουσιαστικά τροπολογίες έχω πάρει, παρόμοιες και οι τρεις, αλλά τρία διαφορετικά αιτήματα. Η πρώτη από των συναδέλφων Άλβαρο και Άουλαν, φιλελεύθεροι. Το δεύτερο από τους σοσιαλιστές Νταρντέν και Γκρέλερ. Αυτές οι δύο τροπολογίες αναφέρονται στο να ξαναρχίσει η συζήτηση για το μέλλον αυτού του Ταμείου. Και σας θυμίζω και τη θέση μου και τη θέση του ΕΛΚ, ότι το μέλλον αυτού του Ταμείου, όπως αρκετά συζητήθηκε στην έκθεση Πόρτας, θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων των προσεχών δημοσιονομικών προοπτικών. Τρίτη τροπολογία, παρόμοια και αυτή με τις άλλες, είμαι υπέρ αυτό που ζητάνε οι συνάδελφοι, οι συνάδελφοι Άλβαρο και Άουλαντ σε φάση οικονομικής κρίσης, λιτότητας, όπως ακούσαμε και χθες. Σωστό είναι η Κομισιόν να βρει νέες budget line, όχι αυτές που κλασικά αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, ελπίζω ότι οι διερμηνείς κατάφεραν να με παρακολουθήσουν. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Τέλεια, κύριε Σιγήτρα. Ο κύριος Άλβαρο. Ευχαριστώ θέμα, πρόεδρε. Οι δικοί μου διερμηνείς εξαιρετικά τα κατάφεραν τουλάχιστον η δική μου. Ευχαριστώ για την εισαγωγή τη εισηγητρία. Σκιώδης για την ομάδα μου και έτσι είναι φυσικό ότι έτσι, σε σχέση με την τροπολογία που ο συνάδελφο έχει καταθέσει και εγώ, διότι σύντομα θα ήθελα να αναφέρω, διότι αναφέρθηκε σε αυτήν η εισηγήτρια. Εμάς θα μας ενδιέφερε μόνο, μια και είδαμε ότι μεταξύ άλλων και οι μεταφορές μεταξύ άλλων από τον τομέα της ανταγωνιστικότητας έγιναν, από εκεί αντλήθηκαν πράγμα που αφορά και πλήττει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι σίγουρα που για το ΕΛΚ είναι εξίσου σημαντικό όπως για μας και για άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες. Και γι' αυτό ο συνάδελφος Χάλλον και εγώ είχαμε καταθέσει την πρώτη τροπολογία. Μήπως δεν θα μπορούσαμε υπό το φως της λογικής χρήσης των κονδυλίων ίσως οι εισηγήτρια και η κοινοβουλευτική της ομάδα να πιστούν να υποστηρίξουν αυτή την τροπολογία, να την υπερψηφίσουν. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστώ, δεν ζητά κανείς άλλο το λόγο, οπότε ε, θέτω προς ψήφιση. Έχουμε τρεις τροπολογίες οι οποίες αναφέρονται στις τρεις εκθέσεις. Euh, Και να δούμε εάν υιοθετείτε μία τροπολογία ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. Έχετε όλη τη λίστα των τροπολογιών στην παράγραφο 5 η τροπολογία 1 του κυρίου Άλβαρο και Χάγκλουγκ. Ο εισηγητής, η εισηγήτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απε, απορρίπτεται. Η τροπολογία 2 του, των κυρίων Ντεντέν και Γκρελιέ. Ποιος είναι ε, υπέρ. Κατά. Επίσης απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Με μια προφορική τροπολογία την οποία έχετε στο κατάλογό σας. Όλοι δηλαδή την έχετε μπροστά σας. Η συγκήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ευχαριστώ. Άρα υπάρχει μία πλειοψηφία υπέρ και ε, εγκρίνεται. Μπορεί λοιπόν να γίνει μία τελική ψηφοφορία ε, για όλες μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Δύο ο κατά δεν υπάρχουν αποχές, άρα και οι τρεις εκθέσεις εγκρίνονται και ευχαριστούμε την εισηγήτρια για την εξαιρετική εργασία και την ταχύτητα με την οποία επέτυχε την ομοφωνία της Επιτροπής Προϋπολογισμού και αποτελεί καλό παράδειγμα για τις επόμενες εκθέσεις και ιδίως για τη συντονία που ελπίζουμε να είναι εξίσου γρήγορη και αποτελεσματική στη συνέχεια. Τώρα έχουμε το σημείο 9 της ημερησίας διατάξεως που αναφέρεται εις τον κανονισμό προσωπικού της ε, υπηρεσίας ε, εξωτερικής δράσης και ε, η εισηγήτρια θα μας πει με τον ίδιο τρόπο σε δύο λεπτά πόσο σκοπεύει να αντιμετωπίσει τις τροπολογίες και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ ψηφίσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης ε, για τον τροποποιημένο κανονισμό προσωπικού σε σχέση με την εισαγωγή και δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Υπηρεσίας. Είναι μια γνωμοδότηση για την ίδια την έκθεση τη Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων επ' αυτού του ιδίου θέματος. Σε μια εβδομάδα θα ψηφιστεί στην Επιτροπή Νομικών. Έχουν κατατεθεί δύο τροπολογίε από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Προστίθενται στις 20 τροπολογίε που είχαν κατατεθεί αρχικά προτείνω επιπλέον τρεις συμβιβαστικές τροπολογίες και τρεις προφορικές τροποποίησεις. Για να υπάρξει διαφάνεια για δημοσιονομικούς λόγους, οι αλλαγές θα πρέπει να περιορίζονται σε εκείνο που είναι εύλογο για την λειτουργία της εξωτερικής υπηρεσίας και όχι τίποτε άλλο. Εξέτασα την πολιτική συμφωνία που ελήφθη τον Ιούνιο και για την διασφάλιση της ε, συμβατότητας των προτάσεων αυτών με αυτέ τι ε, προτάσει. Ωστόσο αξίζει να πούμε ότι σε κάποια θέματα όπω γεωγραφική εκπροσώπηση κτλ. υποστηρίζω του συναδέλφου του ΕΛΚ και Είμαστε σύμφωνοι και ζητούμε να είμαστε σύμφωνοι με τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2010 σε σχέση με απόφαση του Συμβουλίου για την διοργάνωση της εξωτερικής διπλωματικής υπηρεσίας. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. I to be short. Ε, υποσχέθηκα να είμαι σύντομη και ήμουνα και καλύτερα πάμε. Δεν ζητά το λόγο κανείς άλλος και είμαι πανευτυχής. Προτείνω λοιπόν, επειδή όλοι έχετε τον κατάλογο της ψηφοφορίας, θα υπάρξει και μία ε, προφορική ψηφοφορία η οποία θα συζητηθεί και τώρα έχουμε την ε, πρώτη συμβιβαστική τροπολογία α που ετοίμασε η, ε, η συγγήτρια. Ποιος είναι υπέρ. Qui est contre Ah, trois contre, dont ε, ε, Τρεις εκ των οποίων οι πράσινοι. Ε, αποχή υιοθετείται. Το, η τροπολογία Β. Στου στους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Το, η τροπολογία Β κεφαλαίο. Άρα ε, ε, ε, εγκρίνεται. Η συμβιβαστική τροπολογία γάμα κεφαλαίο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν έχουμε αποχές. Άρα εγκρίνεται. Στη συνέχεια έχουμε μία πρώτη ομάδα τροπολογιών που ψηφίζουμε ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στο σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Άρα και τα τρία έχουν καλυφθεί εδώ. Το α κεφαλαίο 1 και 21 έχουν καλυφθεί από την συμβασική τροπολογία μπλοκ 1. Τώρα περνάμε στην πρόταση του κανονισμού. Τροπολογία 10 της συγκήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Χαθήκαμε όλοι, λέγει ο εισηγητής. Είμαστε σελίδα 3, πρόταση για κανονισμό, Proposal for a Regulation, άρθρο 1, σημείο 7, τροπολογία 10 της κυρίας Νέινσκι. Ποιος είναι υπέρ. Στον κατάλογο ψηφοφορίας είναι. Ηλεκτρονικά λοιπόν για ε, την σελίδα 3 του καταλόγου ψηφοφορίας ξεκινάει η ψηφοφορία. Είμαστε 36 στην αίθουσα. Πρέπει να ξυπνήσουμε τους συναδέλφους. Λίγη η ψηφοφορία. 18 υπέρ, 17 κατά εγκρίνεται. Η τροπολογία 28 του κυρίου Γκαλτιέρη. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές, όχι αποχές, εγκρίνεται. Τώρα υπάρχει μια ε, προφορική τροπολογία της κυρίας Νιέσκη που υπάρχει στο δελτίο ψηφοφορίας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία αποχή άρα εγκρίνεται με ευρία πλειοψηφία. Η τροπολογία 12 καλύπτεται από τον μπλοκ 1, η τροπολογία Γ καλύπτεται από τη συμβιβαστική Γ, όπως και οι τροπολογίες 13, 30 και 31 που καλύπτονται από τη συμβιβαστική τροπολογία Γ. Περνάμε τώρα στην ε, ε, προφορική τροπολογία, την οποία ίσως θα μας διαβάσει η συγγήτρια. Αν θέλετε να το διαβάσω, εντάξει. Ήθελα όμως μόνο να πω ότι χθε το βράδυ το ΕΛΚ και οι σοσιαλιστές κατέληξαν σε συμφωνία για την καλύτερη διατύπωση τροπολογίας 29 για την γεωγραφική ισορροπία και έτσι αποφεύγεται η δυνατότητα, η πιθανότητα εσφαλμένης ερμηνείας σαν να εισάγεται ένα σύστημα ποσοστώσεων. Σας διαβάζω τι συμφωνήσαμε, ΕΛΚ και σοσιαλιστές. Θεωρούμε ότι μέσα στο πλαίσιο και τους περιορισμούς του αριθμού S που κατανέμεται βρισκό, ευθυγραμμιζόμαστε σε σχέση με τους στόχους διάδρασής σας στην στελέχωση. Διαγράφουμε το by και λέμε in accordance with, σύμφωνα με, ευθυγραζόμενοι με. Αυτή είναι η μόνη αλλαγή. Καθιστά σαφέστερα το κείμενο και ικανοποιεί σχεδόν όλους. Ευχαριστώ. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι ορισμένοι ε, ορισμένοι ήθελαν να υπάρξει μια γεωγραφική ισορροπία χωρίς να φτάσουν στις ποστοσώσεις ε, αλλά με μία παραπομπή εις ε, την εις, εις την στην γνωστή ρήτρα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξ ονόματο της συναδέλφου Φρανσίσκα λόγω ασθένεια, δεν μπορεί να παραστεί θα να διαβάσω τη δική μα τροπολογία πώ έχει μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020 η στελέχωση για τέτοιου είδους ε, υπαλλήλους θα λαμβάνει υπόψη η πρόσληψή τους ενδεικτικούς στόχους ε, πρόσληψης ε, που θα βρίσκονται ευθυγραμμιζόμενοι με τις κλίδες αναφοράς και μετά σε σχέση με τα κράτη τα οποία υποεκπροσωπούνται θέλουμε να το αναδιατυπώσουμε ως έχει, όπως σας διάβασα. Ευχαριστώ. Madame le Yes, thank you. Uh, Η Παραμένουμε στο δικό μας κείμενο έχει, αυτό προτιμάμε. Υποβάλλω λοιπόν προς ψήφιση την ε, προφορική τροπολογία της εισηγητρίας και διαφορετικά θα ψηφίσουμε την τροπολογία της κυρίας Τρίπελ. Ποιος είναι υπέρ της προφορικής τροπολογίας υπαριθμών 29. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρα καλύπτει και την τροπολογία της Έλγα. Το 14, 15, 16 καλύπτονται από τον μπλοκ 1, το 17 της συγγήτρια. Ποιος είναι υπέρ. Τροπολογία 17. Κατευθείαν λοιπόν η ηλεκτρονική ψηφοφορία ξεκινά και πιστεύω ότι εδώ θα υπάρξει ε, διαφορά. Πάλι η κυρία δεν έχει την ε, κάρτα της ε, ψηφοφορίας οπότε εγώ μπορώ να ψηφίσω. Έχουμε 21 υπέρ, 18 κατά. Είναι πολύ σφιχτά αλλά υιοθετείται. Στο 32 της κυρίας Μπράντερ ε, ο εισηγητής είναι κατά. Κατά. Όλοι οι άλλοι. Μία αποχή. Και άρα απορρίπτεται. Η, ε, η τροπολογία Γκαλτέρη χωρίς αριθμό καλύπτεται από το 17 το οποίο ε, εγκρίναμε ε, οι 18, 19 και 20 καλύπτονται από το μπλοκ 1 καθώς και η, τροπολογία, η πρώτη τροπολογία στην επόμενη σελίδα. Μετά έχουμε... Α, με συγχωρείτε γύρισα πίσω. Μάλλον έκανα όπισθεν. 22. Είναι μία πρόταση του εισηγητή να αλλάξουμε την ε, ε, τοποθέτηση μέσα στο κείμενο ποιος είναι υπέρ. Κατά. Είσαστε κατά. Αποχή. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23 το ίδιο, 24 το ίδιο, 23 και πάλι της ηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 24 της συγγήτριας Υπάρχει μια ελαφρή αλλαγή της, ε, του κειμένου και λέμε representation of certain member state nationals in DG Relex, ηλεκτρονική ψηφοφορία για το 24 και ε, αντικαθιστώ τη συντονία όπως μου το ζήτησε διότι δεν έχει κάρτα. Λίγη η ψηφοφορία. 20 ε, υπέρ, 18 κατά, τσίμα τσίμα περάσαμε. Ε, το... Το 2 καλύπτηκε και από τον μπλοκ το 25 του κυρίου Καλτιάρη υπέρ. Ηλεκτρονικά πάλι. Ξεκινάει η ψηφοφορία ε, και συμμετέχω ο, η αντί για την κυρία Συντονία. Τελειώνει. 22 υπέρ, 16 κατά, άρα η τροπολογία Γκουαλκέρι οθετείται. Οπότε γίνεται η παράγραφος 3β, η τροπολογία 3 προφορική της εισηγητρίας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερα καλύπτεται από τον μπλοκ 1, η τροπολογία 26. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται μόνο οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι κατεψήφισαν. Και ο κύριος Χάρτογκ. Το Β καλύφθηκε, η τροπολογία 5 και 27 καλύπτηκαν από το συμβιβαστική Β, το 6, 7, 8 καλύπτονται από τον μπλοκ 1, η τροπολογία 9 για το εκτιμώντας 17 ποιος είναι υπέρ, η είναι υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία πάλι για την τροπολογία 9. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. 21 υπέρ 18 κατά εγκρίνεται. Και τελειώσαμε. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε τελική ψηφοφορία της εκθήσεως ποιος είναι υπέρ. Κατά. Δύο κατά. Αποχές δεν έχουμε αποχές. Άρα ομοφωνία με μείον δύο και ε, συγχαίρουμε την εισηγήτρια και τους συναδέλφους. Τώρα, αφού Τώρα έχουμε την έκθεση Ανδρέασεν. Έχετε όλοι τον κατάλογο ψηφοφορίας της εκθέσεως της κυρίας Ανδρέασεν. Μπορούμε να προχωρήσουμε κατευθείαν στην... Ε, θέλετε να κάνετε μία δήλωση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα πολλές ευρωπαϊκές χώρες θα απεργήσουν. Και αυτό οφείλεται στα μέτρα λιτότητας που κάποιες ε, κυβερνήσεις προσπάθησαν να εφαρμόσουν. Το να αρνηθεί κανείς ότι πολλές από αυτές τις χώρες είναι οι θεματοφύλακες του συστήματος, του πακέτου διάσωσης θα ήταν μεγάλο σφάλμα. Επίσης μεγάλο σφάλμα θα ήταν να αγνοήσει κανείς ότι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα οφείλεται στην έλλειψη, στην απουσία σεβασμού για το σύμφωνο σταθερότητας έτσι λοιπόν πιστεύω ότι κυρώσεις πρέπει να εφαρμοστούν, να εισαχθούν και πρέπει να είμαστε σοβαροί στην επιβολή κυρώσεων. Ευχαριστώ. Merci, madame. Merci, madame. Très bien. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλο να ζητά το λόγο. Άρα ε, ψηφίζουμε την πρώτη τροπολογία του κυρίου Κοσλόφσκι. Ε, θέλετε το λόγο. Ο κύριος Χάρτουγκ θέλει το λόγο. Θα ήθελα να υποστηρίξω στεναρά την κυρία Ανδρέασεν για την έκθεσή της και είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό να δούμε την πραγματική κατάσταση, τη σημερινή κατάσταση στην Ευρώπη, να υποστηρίξουμε όλα τα μέτρα για την επιβολή κυρώσεων στα κράτη-μέλη που δεν συνεργάζονται και δεν ευθυγραμμίζονται και δεν κάνουν τίποτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι. Τροπολογία 1 του κυρίου Κοσλόφσκι, ε, ποιο είναι υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 Κοσλόφσκι. Η συγγήτρια είναι κατά. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 3 Κοσλόφσκι. Ποιος είναι υπέρ. Η συγγήτρια είναι κατά. Ευχαριστώ. αποχές έχει ε, εγκριθεί. Η τροπολογία 4 η εισηγείται είναι υπέρ. Ποιο είναι κατά. Η Έλγα. Αποχές <clears throat> εγκρίνεται παρά την ε, αντίσταση της ΕΛΓΑ. Ε, τροπολογία 5, εισηγητή ε, κατά, ποιος είναι υπέρ, κατά. Εγκρίνεται επίσης. Τροπολογία 6 προφορική του κυρίου Κοσλόφσκι έχετε το κείμενο μπροστά σας η συγγήτρια είναι υπέρ ποιος είναι υπέρ κατά μία κατά αποχές δεν υπάρχει αποχές εγκρίνεται Επτά, Κοσλόφσκι η συγκίτρια είναι υπέρ ποιος είναι κατά αποχές επίσης εγκρίνεται ε, νέα η συγκίτρια κατά κατά 11. Εγκρίνεται. 8 της κυρίας Χολμάγερ αποσύρεται. 10 Κοσλόφσκι. Προφορική τροπολογία έχετε μπροστά σας στο κείμενο. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. οι σοσιαλιστές απέχουν αλλά εγκρίθηκε. Περνάμε στις τροπολογίες τρίπελ. Μπορώ να τις παρουσιάσω μαζί, τις τρεις της Έλγα, όχι. Λοιπόν, 11 Έλγα τρίπελ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Η εισηγήτρια είναι κατά. Υπέρ. Τι κάνει το ΕΛΚ εκεί. Ελεκτρονική ψηφοφορία στο 12 για να ξυπνήσει το ΕΛΚ. Γιατί έχουμε δύο συντονιστές, αν κοιμούνται και οι δύο. Λοιπόν, λίγη ψηφοφορία. Ένα συνάδελφος ακόμη κοιμάται. 14 υπέρ, 24 κατά, απορρίπτεται η τροπολογία 12. 13 της Χέλγα. ηλεκτρονική ψηφοφορία και πάλι. Δύο συνάδελφοι κοιμώντουσαν αλλά ξύπνησαν όλοι. 25 κατά, 13 υπέρ, μία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται και μου λέγουν ότι πλέον δεν θα χρειαστεί να ψηφίζω διότι μετά από 48 ώρες κατάφερε η συγγήτριά μας να βρει μία κάρτα ψηφοφορίας. Όλοι προοδεύουμε. Τώρα που βρισκόμαστε, 12, 13, έχω χάσει το λογαριασμό. 14 Κοσλόφσκι, η συγγήτρια είναι υπέρ, υπέρ. Κατά. Αποχές, δύο αποχές. 14 εγκρίνεται. 15 ε, Κοσλόφσκι εισηγητής είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία αποχή. Εγκρίνεται. 16. Μία τροπολογία Κοσλόσχη με μία μακριά προφορική τροπολογία των σοσιαλιστών. Ο εισηγητής είναι κατά. Έχετε μπροστά στο κείμενο ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ο εισηγητής και τρεις ακόμη. Ποιος απέχει εγκρίνεται. 17 Κοσλόφσκι. Ο εισηγήτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 Κοσλόφσκι. Η εισηγήτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Υπάρχει μία μικρή πλειοψηφία. Αποχές υπάρχει μία συνήθις πλειοψηφία αλλά ε, ε υιοθετείται. Η 19 Χολμάιερ δεν έχει ε, αποσυρθεί, είναι ε, ίση με την 18 του Κοσλόφσκι. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές. Επίσης εγκρίνεται παρό, παρά την αντίσταση της εισηγητρίας. Τώρα λοιπόν ο, ψηφίζουμε την έκθεση κατά δύο αποχές. Άρα η έκθεση, μάλλον η γνωμοδότηση εγκρίνεται και ευχαριστώ την εισηγήτρια που έκανε μια πολύ ποιοτική εργασία. Άρα, τώρα ολοκληρώσαμε αυτές τις ψηφοφορίες, αλλά πριν αρχίσουμε επί του προϋπολογισμού, και όσο ζεστάνει η συντονία την κάρτα ψηφοφορίας που μόλις έλαβε, έχουμε μεταφορές να κάνουμε. Εμβάσματα. Ξεκινάμε λοιπόν με τα εμβάσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα το 14, 15 και 20 που αναφέρονται εις ε, τις ε, μετακινήσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο της Προσαρμογής της Παγκοσμιοποίησης, δηλαδή στην έκθεση που υιοθετήσαμε της κυρίας Ματέρα, οπότε φαντάζομαι ότι ο κύριος Σούργιαν ο εισηγητής είναι υπέρ των τριών αυτών ε, μεταφορών. Δεν μιλάει, αλλά επειδή κουνάει το κεφάλι του αντιλαμβάνεστε ότι συμφωνεί. Θέλει όμως τώρα να μιλήσει ο Λάσλο. Του δίνω το λόγο. Μάλλον είπε ναι. Από κοινού 14, 15 και 20. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν έχουμε αποχές. Άρα οι τρεις αυτές ε, μεταφορές εγκρίνονται. info 1. Info 1. Και υπάρχει και info 2. Μπορούμε να τα ψηφίσουμε μαζί. Κύριε Πρόεδρε, καλό θα ήτανε να ε, ε, παρουσιάσουμε μια επισκόπηση αυτών των μεταφορών οπότε θα έλεγα τουλάχιστον εγώ ε, να ψηφίσουμε όλες τις μεταφορές μαζί διότι εγώ τις στηρίζω. Άρα από κοινού για το info 1, info 2, solvit, tsc 44 εγώ αυτά έχω όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ίγκε θέλει να λάβει το λόγο. Μια ερώτηση να κάνω, μια ερώτηση. <clears throat> Στον τύπο για αυτή την ε, επιχείρηση, για αυτήν την εταιρεία, για μια τηλεοπτική, ένα τηλεοπτικό συνεδρίο. Θα ήθελα να ξέρω αν ο λόγος για αυτή τη μεταφορά εντάσσεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο αυτής τη υπόθεση. Ήταν αυτό το θέμα της επικοινωνίας, μεταφορά για θέματα επικοινωνίας, στον τομέα της επικοινωνίας. Ο αντιπρόεδρος Αλβαρό μας λέει ότι δεν πρόκειται γι' αυτό. Όχι, δεν εντάσσεται στον τομέα της επικοινωνίας, κυρία, αλλά στον τομέα 3 θα εντασσόταν που στη συνέχεια θα ψηφίσουμε αλλά έχουμε συμφωνήσει με πλευρά εσύ ότι θα υπάρξει μια προφορική τροποποίηση, αλλά δεν αφορά αυτή τη μεταφορά. Ή τα κονδύλια για την επικοινωνία δεν εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο αυτής της μεταφοράς. Bien. Donc, on traite pas ça maintenant, mais rendez-vous est pris pour... Λοιπόν, δεν θα το ε, λύσουμε τώρα, αλλά κάποια στιγμή στο μέλλον. Ποιος είναι υπέρ ο μπλοκ των ε, μεταφορών. Μήπως ο σοσιαλιστής συντονιστής μπορεί να μας πει τι σκέφτεται υπέρ, κατά. Αποχές, μία αποχή εγκρίνονται. οι άλλες μεταφορές στη, στα άλλα θέματα δεν είναι έτοιμος ο εισηγητής, οπότε δεν θα ψηφιστούν τώρα. Τώρα, ολοκληρώσαμε όλες τις ψηφοφορίες για θέματα εκτός προπολογισμού και μπορούμε να επανέλθουμε στον προπολογισμό. Προβλέψαμε εχθές να ξεκινήσουμε τις ε, ψηφοφορίες σήμερα το πρωί. Ε, ε ξεκινάμε με 20 λεπτά καθυστέρηση και θα ψηφίσουμε την κατηγορία 1α. Voilà. Est-ce que tout le monde a, euh, est en position Voilà, j'espère que je suis... Κάθεστε όλοι. Ελπίζω ότι και εγώ είμαι έτοιμο, αλλά δεν είμαι και βέβαιο. Λοιπόν, μιλάμε για την ε, αηφόρο ανάπτυξη, sustainable growth. Αυτό είναι ο τίτλος των εργασιών μας σήμερα. Μήπως η συγγήτρια θέλει να κάνει κάποια δήλωση πριν την ψηφοφορία στο 1α ή όχι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω την πολύ δύσκολη κατάσταση που έχουμε στο κεφάλαιο 1α. Για να υπενθυμίσω, υπό αυτό αυτόν τον τίτλο υπάρχει μια σειρά πολύ σημαντικών προτεραιοτήτων ως κονδύλια για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προγράμματα έρευνας, για παράδειγμα. Προγράμματα που συνδέονται με την εκπαίδευση, παιδεία, κατάρτιση, κινητικότητα στην εκπαίδευση και παιδεία. Και ήδη τα κονδύλια, οι πόροι που προβλέπονται από το MFF έχουν εξαντληθεί. Το περιθώριο ελιγμών μας σε αυτή την κατηγορία, σε αυτόν τον τίτλο είναι πολύ περιορισμένο. Και αυτό που έκανε το Συμβούλιο είναι σημαντικές περιστολές, σημαντικοί περιορισμοί σε σημαντικά κονδύλια. Ένα παράδειγμα να δώσω σε σχέση με τις εκτελεστικές υπηρεσίες που θα υλοποιήσουν το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη. Η κυριότερη πρότασή μου για αυτό το τον τίτλο είναι να αποκατασταθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό το σχέδιο προϋπολογισμού. Είμαι πεισμένη ότι χρειάζονται αυτές οι δεσμεύσεις πιστώσεων υποχρεώσεων για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα όπως προβλεπόταν από την νομοθετική βάση. Να επανέλθουμε στο προσχέδιο προϋπολογισμού λοιπόν, αλλά είναι εξίσου σημαντική η διάσταση σημαντικά κονδύλια να ενταχθούν σε αυτό το κατάλογο σε αυτόν τον τίτλο. Να υπενθυμίσω αν επιτρέπετε ότι εχθές ψηφίσαμε μια οριζόντια τροπολογία από πλευρά εισηγητού σε κάποιες από τις προτεραιότητες για τα κονδύλια που θα τα ξαναδούμε όταν πρόκειται να έρθουμε και ψηφίσουμε για αυτά. Υπάρχουν αρκετά λοιπόν, αρκετές αυξήσεις που προτείνονται από, μια, από τις εξειδικευμένες κοινοβουλευτικές επιτροπές και πιστεύω ότι υποστηρίζουμε αυτές τις συστάσεις. Αν όμως υποστηρίζουμε αυτές τις σημαντικές ε, επί της ουσίας αυξήσεις, αντιμετωπίζουμε την κατάσταση να έχουμε 29 εκατομμύρια ευρώ που θα ξεπεράσουμε την οροφή κατά αυτό το ποσό, 29 εκατομμύρια ευρώ. Η πρόταση που συζητείτε με τους συντονιστές είναι να μπορέσουμε αυτό το κονδύλιο να το αντισταθμίσουμε, να το αντισταθμίσουμε με περικοπή στο πρόγραμμα ITER. Ουσιαστικά παραμένουμε έτσι μέσα στο πλαίσιο του περιθωρίου, μέσα στην οροφή. Αυτή είναι η πρόταση για την αύξηση των κυριότερων γραμμών που επιθυμούμε, διαβίου εκπαίδευση, lifelong learning, πρόγραμμα SIT κτλ και να αντισταθμιστούν αυτές οι αυξήσεις με μια περικοπή στα κονδύλια ΙΤΕΡ. Και μια και έχω τον λόγο αν επιτρέπετε. Η ιδέα είναι να ψηφίσουμε κονδύλιο ανά κονδύλιο στον τίτλο αυτό και εγώ θα συστήσω ακολουθώντας την φιλοσοφία που μας εμπνέει και σας εξέθεσα θα είμαι υπέρ και θα σας εξηγήσω να είμαστε υπέρ ή κατά κάθε τροπολογίας ανάλογα. Ωστόσο είναι σημαντικό ότι υπενθυμίζω Κάποιοι από εσά θα έχουν ίσως αμφιβολίες για τις περικοπές των κονδυλίων ίτερ. Αν υποστηρίζετε όλες τις αυξήσεις στα κονδύλια που προτείνουμε, να θυμόμαστε ότι 30 εκατομμύρια ξεπερνάμε την οροφή. Αν δεν είσαστε υπέρ της ε, περικοπής των κονδυλίων ίτερ, τότε αυτό θα σημαίνει ότι ξεπερνάμε την οροφή ούτως ή άλλως κάτι το οποίο δεν υποστηρίζω με κανένα τρόπο και έτσι γι' αυτό τον λόγο υποστήριξα αυτή τη θέση. Συνεχίζοντας τώρα για το μηχανισμό ψηφοφορίας προτείνω όταν έρθει η ώρα να ψηφίσουμε για το κονδύλιο ΙΤΕΡ να ψηφίσουμε την τροπολογία που ε, πάει για την ε, διαγραφή, πάει πιο μακριά, για τη διαγραφή της, ε, του κονδυλίου, πράγμα το οποίο δεν υποστηρίζω και για το ΙΤΕΡ προτείνω να ψηφίσουμε αύριο, Πρόεδρε όταν θα έχουμε το σύνολο, συνολικό ποσό υπόψη για το οποίο θα ψηφίσουμε. Ψηφίζοντας κονδύλιο ανακονδύλιο μπορούμε τη συμφωνία για την περικοπή ίτερ να την προσαρμόσουμε αντίστοιχα. Αν θέλετε και τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάποια συμφωνία από πλευρά συντονιστών εκτιμόμενο ποσό 50 εκατομμυρίων στον τίτλο στην κατηγορία 1α τότε θα πρέπει να έχουμε μια περικοπή 45 εκατομμυρίων του κονδυλίου ΙΤΕΡ αντίστοιχα. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ζητήσω να υποστηρίξετε αυτή την στρατηγική που ακολουθούμε και σας προτείνουμε. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, έχω δύο τεχνικής ε, φύσης παρατηρήσεις. Κάποιοι από εσάς έχουν καταθέσει τροπολογίες που αναφέρουν κάποια ποσά τα οποία θα έπρεπε να διασφαλιστούν για τη χρηματοδότηση της μιας ή άλλης δράσης. Αυτός είναι ένας τρόπος προκαθορισμού κονδυλίων, πράγμα που δεν επιτρέπεται από τον δημοσιονομικό κανονισμό. Η πρότασή μου λοιπόν είναι, σε περίπτωση έγκρισης αυτών των τροπολογιών, να αλλάξουμε κάθε φορά αυτό, αυτό το earmarking, τον προκαθορισμό, να πούμε ότι πρόκειται για appropriations, για πιστώσεις ε, πληρωμών και για τις προπαρασκευαστικές δράσεις και ένα κατάλογό τους. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταφέρει να καταλήξουμε σε μια λύση πακέτο μεταξύ των συντονιστών. Εργαζόμαστε για να πετύχουμε αυτή την λύση, επίλυση του προβλήματος. Προτείνω να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε για μια λύση πακέτο. Ω εισηγήτρια όμω είδα και παρατήρησα ότι πολλά από τα πιλωτικά σχέδια και προπαρασκευαστικά μέτρα έχουν σημαντικά μέτρα ε, και μηνύματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται τα οποία όμω δεν μπορούν όλα να χρηματοδοτηθούν, μια και δεν έχουμε κονδύλια πόρου. Κάποια όμω από τα μηνύματα ή, ή τι παρατηρήσει που συμπεριλαμβάνονται πρέπει να ενταχθούν στο αντίστοιχο κονδύλιο. Προτείνω ω εξή να ψηφίσουμε για αυτέ τι παρατηρήσει. Αύριο θα πάρετε αυτές τις παρατηρήσεις, αυτά τα σχόλια που θα διηθήσω εγώ, θα φιλτράρω από τα πιλωτικά προγράμματα και πιλωτικές δράσεις και θα προτείνω να ενταχθούν στα επιμέρους κονδύλια. Και θα έχετε αυτές τις προτάσεις από πλευράς μου αύριο. Ευχαριστώ. Σε ένα σημείο θα ήθελα να τονίσω κάτι. Ο δημοσιονομικός κανονισμός δεν μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό που συνηθίζαμε να κάνουμε. Δηλαδή έχουμε σχόλια και να ζητάμε η πίστοση που ανοίγουμε να δοθεί σε τέτοιο ποσό, στο α ποσό για αυτή τη δράση, σε β ποσό για αυτή τη δράση, το earmarking που λέμε. Αυτό το δικαίωμα δεν το έχουμε πια. Αντίθετα, μπορούμε να κάνουμε υποδείξεις, προτάσεις χωρίς νούμερο στα σχόλια. Μπορούμε να πούμε ένα τμήμα αυτού, της πίστοσης μπορεί να πάει εκεί. Φέρμα, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τη Συντόνια. Πράγματι ε, κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να βρει πολιτική λύση για το 1α, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να δεχθούμε την πολιτική γραμμή της εισηγήτρια. Είναι κάπως υπερβολικός που να δεχτεί το μήνυμα λιτότητας δεν θεωρούμε ότι η κρίση θα πρέπει να είναι τόσο πολύ σε βάρος σημαντικών προγραμμάτων βέβαια. Αναλαμβάνουμε και εμείς την ευθύνη για τη δύσκολη κατάσταση που σημαίνει ότι δεν δεχόμαστε όλες τις αυξήσεις αλλά θα ψηφίσουμε υπέρ περίπου 25 γραμμών που θεωρούμε σημαντικές προτεραιότητες και ο τρόπος της ψηφοφορίας μας θα κριθεί από το τι συζητήθηκε και στην Ήτρε και σε άλλες επιτροπές. Έχουμε διαφορετική πολιτική γραμμή. Συμφωνούμε όμως με τη Συντόνια για την διαδικασία ψηφοφορία. Να ψηφίσουμε με τη βάση το voting list και στο τέλος να ψηφίσουμε τη γραμμή για το ITER, την buffer line να την πούμε, σαν γραμμή που θα παίξει, παίξει το ρόλο από σβεστήρα. Πρόεδρος, σε ευχαριστώ Γκέραν για το ότι με διευκολύνεις ως πρόεδρο στην οργάνωση της ψηφοφορίας. Το αποτέλεσμα βέβαια εξαρτάται από εσά. Το οργανωτικό όμω σκέλος εξαρτάται και από το Προεδρείο. Σαλβατόρ Γκαρίγκα. Ναι, Πρόεδρε. Θέλω να επιμείνω και να εμείνω στην σύσταση που υπέβαλε ως πρόταση η συγγήτρια που αφορά την ευαίσθητη κατάσταση σε αυτή την κατηγορία 1α στην οποία ως συντονιστές προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε μια κοινή συμφωνία και τελικά δεν ήταν εφικτό, δεν ήταν δυνατό να την πετύχουμε αυτή τη συμφωνία. Θέλω να υπενθυμίσω ότι αυτές οι πρόσθετες τροπολογίες που ζητεί η σοσιαλιστική ομάδα και καταθέτει σημαίνουν εκατομμύρια ευρώ που θα προσθεθούν επιπλέον σε αυτή την κατηγορία 1α και θα πρέπει να προέλθουν από επιπρόσθετες περικοπές του προγράμματος Ίτερ Πιστεύω ότι δεν είναι μια δημοσιονομική πρακτική που να είναι αρκετά σοβαρή αυτή το να θεωρηθεί αυτό το πρόγραμμα ITER ως μια εικονική γραμμή από την οποία μπορούμε να αντλούμε κονδύλια κατά το δοκούν συνεχώς ώστε να υλοποιηθούν άλλες προτεραιότητες και γι' αυτό σε σχέση με αυτή την πρόταση των σοσιαλιστών παρακαλώ να λάβουν υπόψη τις δυσκολίες αυτής της κατηγορίας και τις ανάγκες να βρεθεί χρηματοδότηση και για το πρόγραμμα ITER και γι' αυτό να δεχθούμε την πρόταση που έκανε η Συντόνια που νομίζω ότι επιτρέπει να υλοποιήσουμε τους στόχους της λιτότητας και της προτεραιότητας του Κοινοβουλίου και την πραγματικότητα την πολιτική την οποία θα αντιμετωπίσουμε όταν θα έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη ανάγνωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα για τους σοσιαλιστές συναδέλφους ε, ήθελα να πω ότι κάπως δεν έχουν ίσως συνειδητοποιήσει ποιες θα είναι οι εξοικονομήσεις ε, για να δούμε πόσοι άνθρωποι θα κατέβουν στους δρόμους σήμερα ώστε να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους. 45% των νέων είναι άνεργοι σήμερα. Κατά τούτο αυτό θα έπρεπε να είναι ένα μήνυμα για τους σοσιαλιστές, να καταλάβουν ότι πρέπει να υπάρξουν εξοικονομήσεις. Δεν πρόκειται για χρήματα μόνο, αλλά πρόκειται για την ύπαρξη, την επιβίωση των ανθρώπων, αυτό το πούμε κάθετα. Δεν έχω άλλα σχόλια, αρχίζουμε την ψηφοφορία. Sustainable Growth είναι η σελίδα 3 στο αγγλικό κείμενο τροπολογία 820 ε, εισηγήτρια κατά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 721 Δεν θέλω να καθυστερήσω την ψηφοφορία. Αλλά είναι σημαντική αυτή για το μηχανισμό χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Δεν είναι η μέση γραμμή του προπολογισμού. Εσείς και πρόεδρε μιλήσατε για τη σημασία να βρεθεί λύση στο πρόβλημα αυτό. Ελπίζω να ψηφίσουμε τη γραμμή αυτή όχι για τον προπολογισμό του 2011, και να έχουμε ένα πολιτικό εργαλείο για να μπορούμε να το συζητάμε το θέμα αυτό. Η συγκίτρια ήταν πριν, τώρα άλλαξε γνώμη. 721 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψήφος. Nous sommes 40 présents, 38 votants. Réveillez-vous. Il y a deux votants qui dorment. Δύο ε, συνάδελφοι κοιμώνται, δεν ψηφίσανε. Ένα ψήφισε, άλλο ένα κοιμάται. Πέρα. Κάποιο δεν ξύπνησε. Λοιπόν, 20 κατά, 19 υπέρ απορρίπτεται. 137. Η συγκίτρια είναι κατά. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 317. Εισηγήτρια υπέρ υπέρ. Κατά ηλεκτρονική ψήφος. Ηλεκτρονική το 317. Το βρήκες. Το βρήκες. Το Εξακολουθεί κάποιος και κοιμάται. Α, ξύπνησε. Ξύπνησε. Είναι εξτρέμις. Απορρίπτεται με 21-19 και μία εποχή 42-55. Η είναι κατά. Ποιος euh. Θεαματική αντιστροφή της κατάστασης. Η είναι υπέρ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται λοιπόν η 42-55 47 Ερενάζερ η συγκήτρια είναι κατά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Nous, nous rencontrons de nouveaux amendements de M. Ehrenhauser qui veut diminuer de 10% toutes les lignes. Υπάρχει μια πρόταση για μείωση κατά 10% όλων των γραμμών. Μπορεί να υπάρχουν βέβαια διαφορετικέ τροπολογίε του κ. Ερενχάουζερ, αυτέ θα τι ψηφίζουμε. Διαφορετικά θα εφαρμόζουμε την νομολογία Ερενχάουζερ για να μην ψηφίσουμε. Επόμενη σελίδα. Όλη η επόμενη σελίδα 4 στα αγγλικά καλύπτεται. Σελίδα 68 και 69 το ιδιο 4622 46-22 Ερενχάουζερ. Κλασική νομολογία Ερενχάουζερ θεωρούμε ότι απορρίπτεται. 427. Μας λένε ότι έχουμε χωρική ψηφορία les chiffres et le commentaire. Sur les chiffres, le rapporteur... Για το νούμερο η συγκίτρια συμφωνεί. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ευχαριστώ. Το νούμερο του 427 εγκρίνεται. Τώρα τα σχόλια του 427. Η συγκίτρια είναι υπέρ. Το ΕΛΚ κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πάλι κοιμώνται δύο. Πέρασε. Απορρίπτεται με 19-18. Τα σχόλια απορρίπτονται. Έχουμε τα νούμερα, δεν ξέρουμε σε τι χρησιμεύουν. Όλες οι άλλες τροπολογίες μέχρι το τέρος της σελίδας 5 καλύπτονται. Γυρίζω σελίδα. 729. Δεν ξέρω η συγκίτρια τι λέει, είναι κατά. Ψηφίζουμε. 729, υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ. Μια μικρή πλειοψηφία κατά και αποχές υπέρ. Ε, η 729 αποσύρεται 41-24 καταπίπτει. Η υπόλοιπη σελίδα καλύπτεται. Όχι, λάθος. Δεν καλύπτεται, αλλά δεν το ψηφίζουμε γιατί είναι πιλωτικά προγράμματα. Το ίδιο και τη σελίδα 7 στα αγγλικά. Πιλωτικά προγράμματα. Το ίδιο για τη σελίδα 8. Σελίδα 9. Το πρώτο τμήμα το ίδιο, πιλωτικά προγράμματα, αύριο αυτό. 02-02-15 το διαστημικό πρόγραμμα G-MES τροπολογία Χάρτονγκ 41-26 για διαγραφή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 138 και 694 ταυτόσιμες. Η συγκίτρια είναι κατά. Ψηφίζουμε υπέρ. Είναι 138 υπέρ. Ή ηλεκτρονικά η 138. Βιαστείτε, ψηφίστε. Πολύ ωραία. Όλοι είναι ξύπνοι. 24 κατά 14 πέρα απορρίπτεται. 33 εισηγήτρια είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Καμία εγκρίνεται. 34. Εισηγήτρια υπέρ. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. εγκρίνεται. Διαστημική έρευνα για το διάστημα. 41-27 χάρτων υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 73. Εισηγήτρια υπέρ. Υπέρ. 4287 87 λέει είναι ταυτόσιμη λέει ο πρόεδρος. Η συγγήτρια είναι υπέρ υπέρ. Κατά. Αποχές. Αυτές οι δύο ταυτόσιμες τροπολογίες εγκρίνονται. 640. Ψηφίζουμε μόνο τα σχόλια. 640. Λάθος, συγγνώμη, έκανα λάθος. η Νομίζω πάτε πολύ γρήγορα, Πρόεδρε, στην ψηφοφορία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Υπερβολικά γρήγορα πάω, ναι. Την 42-87 ψηφίσαμε τώρα, την 41-27 θα έπρεπε να ψηφίσουμε. Στο 04-02 για την έρευνα, για την ανάπτυξη. Για την ανάπτυξη στην έρευνα. Ζητώ συγγνώμη. Επειδή τα νούμερα των τροπολογιών είναι τα ίδια, σχεδόν έκανα λάθος. Όχι τα ίδια, είναι τα ίδια. Και διέγραψα οποιαδήποτε ασφάλεια όσον αφορά την έρευνα. Υπερβολικό αυτό. Έχουμε λοιπόν μία τροπολογία Χάρτονγκ. 41-27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ευχαριστώ. Τώρα σας προτείνω για τις τροπολογίες Χάρτονγκ, γιατί έχουμε και άλλες, και διαγραφή να θεωρούμε ότι υπάρχει πλειοψηφία κατά. Αντίθετα, αν υπάρχουν άλλε άλλες τροπολογίες θα τις ψηφίζουμε. 73. Της Επιτροπής Έρευνας. Η συγγήτρια υπέρ, υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 4286 καλύπτεται. Αντιψηφίζουμε τώρα ξανά την 640 που αφορά τα σχόλια. Η συγκίτρια είναι υπέρ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Πλειοψηφία υπέρ. Εγκρίνουν τα σχόλια. 4127. Χάρτον. Νομολογία χάρτον. 41-28. Παρατρέχω μου φαίνεται λέει ο πρόεδρος. Για να δούμε. Συγγνώμη. Πολύ συγγνώμη είναι τυπωμένα αντίθετα πέρα τη σελίδα 10 στη 12. Mais peut-être que vous êtes dans la même situation que moi, je ne sais pas. Donc, en haut de la page 11. Στο πρώτο μέρο τη σελίδα 11, η United Satellite Programs, Έγνος και Γκαγιλαίο. 41-28 νομολογία Χάρτον. Πρέπει να ψηφίσουμε την 74. Εισηγήτρια κατά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 74. Ο ισχυρό αντιπρόεδρος Ντεάν θα ψηφίσει. Όχι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Απορρίπτεται. Και 695 καταπίπτει. 41-28, 75-44-71 καλύπτονται. Η 41-28 της GNSS νομολογία χάρτων και το κάτω μέρος σελίδας καλύπτεται. Σελίδα 12. Έχουμε τροπολογίες Ehrenhauser ή συνήθες, μείωση κατά 10% πλειοψηφία κατά. Σελίδα 13. 433 νομολογία χάρτων. 450 ψηφίζουμε. η Εισηγήτρια υπέρ. Α, χωριστή ψηφοφορία εδώ, δύο τμήματα. Πρώτα το νούμερο. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ του νούμερου. Ποιος είναι κατά το νούμερο. Τρεις το νούμερο της 450 μένουν. Τα σχόλια του 450, η συγγήτρια υπέρ. Ηλεκτρονικά. ...39 άτομα, 22 κατά. Και εδώ έχουμε τα νούμερα χωρίς σχόλιο, δεν ξέρουμε πού προορίζονται. 306 καταπίπτει, 77 καλύπτεται, 41-33 νομολογία χάτων, 451. Χωριστή ψηφοφορία. Πρώτα νούμερο. Η συγγήτρια υπέρ, υπέρ. Κατά. Πολύ. Αλλά οι περισσότεροι είναι υπέρ. εγκρίνει το νούμερο. Το σχόλιο, η συγγήτρια είναι υπέρ ηλεκτρονική ψήφος. 39 26 κατά, 13 υπέρ. Και εδώ έχουμε μια γραμμή χωρίς να ξέρουμε σε τι θα τη χρησιμοποιήσουμε. Τα υπόλοιπα της σελίδα καλύπτονται. Σελίδα 14. 41-33 χάρτον. 823 κατά. Υπέρ. Κανείς κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. απορίπετα Έρεν Χάζερ διαφορετική όμως. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ αποχές ομόφωνα κατά. 452. Η συγκίτρια υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 701. Το 42-19 είναι ταυτόσιμοι. 701 πρέπει να ψηφιστεί. Είναι μόνο σχόλια. Η συγκίτρια είναι κατά. Ψηφίζουμε. Ηλεκτρονικά. Τα σχόλια της 701. Πέρας. Ψηφίστε μπράβο πολύ γρήγορα. 21-16. Απορρίπτεται. Και εδώ χρήματα χωρίς να ξέρουμε τι θα τα κάνουμε. 41, 33, 46, 18 κλασικές απορρίπτονται 453 η συγγήτρια υπέρ μου λένε ότι η συγγήτρια είναι υπέρ ναι είναι υπέρ υπέρ κατά πολύ αλλά όχι πλειοψηφία αποχές εγκρίνεται όλες οι άλλες καλύπτονται. Τελειώσαμε τη σελίδα 15 αγγλικά. Σελίδα 16. Τροπολογία 470 σελίδα υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 174 η συγκέντρια είναι υπέρ. Επιτροπή γυναικών, ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 471 καλύπτεται. 612. Αφορά μόνο τα σχόλια. Η συγκέντρια είναι κατά. Όχι, είναι υπέρ. Είναι υπέρ. Ψηφίζουμε υπέρ κατά ένας καμία αποχή εγκρίνεται η άλλη είναι ταυτόσιμη στο τέλος πιλωτικά προγράμματα αύριο αυτά όλη η σελίδα 17 πιλωτικά οι προτεραιότητες το ίδιο για τη σελίδα 18 σελίδα 19. Κλασική χάρτον απορρίπτεται. 824. Εισηγήτρια κατά. Υπέρ. Κανεί κατά. αποχέ. Έγινε σκόνη αυτή η τροπολογία. 4.59. Εισηγήτρια είναι υπέρ. Κατά. αποχές πλειοψηφία υπέρ 460 μόνο τα σχόλια η υπέρ υπέρ ευχαριστώ κατά αποχές εγκρίνουν τα σχόλια εδώ ξέρουμε τι θα τα κάνουμε τα λεφτά αυτά 613. Informal carers, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, τέλο πάντων, τα σχόλια μόνο υπέρ, κατά αποχές 4335 43-35 ταυτόσημη. Κοινωνική προστασία και συμμετοχή. 41-34 απορρίπτεται εισηγήτρια κατά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 461 εισηγήτρια υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 472 καλύπτεται 614 Informal carriers πάλι ψηφίζουμε. Η συγκίτρια είναι υπέρ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται με μία αποχή. Η επόμενη καλύπτεται. Σελίδα 20. Working conditions. 826. Η κατά υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 462 εισηγήτρια υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οι άλλες καλύπτονται με εξαίρεση του informal carers να μου εξηγούσε κάποιος τι σημαίνει 615 η εισηγήτρια είναι υπέρ υπέρ κατά αποχές ομόφωνα δεκτή για τους informal carers 43-37 καλύπτεται anti-discrimination 41-34 νομολογία χάρτων 8-27 εισηγήτρια κατά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 597 στους πράσινους υπέρ η σύγκριτα είναι κατά υπέρ η πράσινη κατά όλοι οι άλλοι αποχές συντρίφτηκε δηλώσει αυτή 463 μόνο τα σχόλια η συγκίτρια υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 616. Σχόλια. Η υπέρ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Η επόμενη είναι ταυτόσιμη. Καλύπτει. Gender Equality. 41-34 κλασική χαρτον 828 Η κατά υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτε 599 εισηγήτρια κατά υπέρ κατά όλοι αποχές απορρίπτε 617 informal carriers πάλι εισηγήτρια υπέρ υπέρ κατά αποχές όλοι είναι υπέρ ναι. δεκτή 590 των πρασίνων εισηγήτρια κατά υπέρ Η ηλεκτρονική ψήφος, γιατί εδώ η πράσινη βρήκαν συμμάχος. Ο ένας από όλους δεν ψήφισε. 23-15 απορρίπτεται. Support for Implementation 474. Δική μας Επιτροπή Εισηγήτρια υπέρ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 42-41 πιλωτικό. 41-34 Χάρτον απορρίπτεται. Γύριζε σελίδα. 22. 41-34. Αλλά στο Institute for Gender Equality. Χάρτον. Κλασική. Απορρίπτεται. Ό,τι αφορά την υπηρεσία για την βελτίωση των συνθηκών εργασία. καλύπτονται. Πάμε στο Κατηγορία 2, 42-34 του κ. Λούκας, απορρίπτε Και ένα 46-61 του κ. Αρχάζου για το προφηματικό Αυτή την Η συγκήτρια είναι κατά. 46-61. Η συγκήτρια. Αυτή η τροπολογία καλύπτεται από την οριζόντια τροπολογία για το έλλειμμα. Εγώ Είμαι στη γραμμή 04040302. Συμφωνούμε. Η 4661 καλύπτεται λέτε. Μάλιστα. Δεν ψηφίζουμε. Η επόμενη γραμμή. European Agency for Safety and Health at Work. Άλλη υπηρεσία αυτή. Όλα αυτά καλύπτονται. Μου λέει η επικεφαλής των υπηρεσιών που κάθεται στα αριστερά μου. Η 46-60 καλύπτεται. Ναι. 477. Αυτή δεν καλύπτεται. Ψηφίζουμε. Συγγήτρια υπέρ, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πιλωτικά προγράμματα. Προχωρούμε, γυρίζω σελίδα. 24. European Year for Combating Poverty and Social Exclusion 478 εισηγήτρια υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε οι άλλες δύο ταυτόσιμες καταπίπτουν. πιλωτικά πάμε στο κάτω μέρος European Microfinance Facility Χάρτον 34. απορρίπτεται Επόμενη σελίδα πιλωτικά. Μπορούμε να γυρίσουμε τη σελίδα. Σελίδα 26 πάνω πιλωτικό. Αυτό για αργότερα. Και ερχόμαστε στο EGF που η Μπάρμπαρα την ενδιαφέρει ιδιαίτερα αλλά δεν είναι στην αίθουσα. 628. Η συγγήτρια κατά. Υπέρ. Κάτι μου λέει η Υπήρχε έτοιμα σε τμήματα ψηφοφορίας. Πρέπει να ψηφίσουμε τις παρατηρήσεις, πιστεύω. Ναι, δεν είναι προμεμόρια, δεν έχει νούμερο. Ναι, αλλά μόνο τα σχόλια της παρατηρήσεις θα πρέπει να ψηφίσουμε μόνο. Και την πιο πέρα τροπολογία για τα ποσά που ξεκινά με την τροπολογία 829 για την τροπολογία 628 θα έπρεπε μόνο τις παρατηρήσεις να ψηφίσουμε και μετά να περάσουμε και να ψηφίσουμε την 829 που είναι η μεγαλύτερη πρόταση που έχουμε για ποσά. Ευχαριστώ. Vous, autrement dit... Δηλαδή λέτε να ψηφίσουμε τα σχόλια πριν τα νούμερα. Πριν από τα νούμερα. Περίεργο αυτό. Η κυρία Γένσεν. Συμφωνώ με τη Συντόνια. Πρέπει πρώτα να, πρέπει να ψηφίσουμε ξεχωριστά παρατηρήσεις και ποσά ξεχωριστά. Θα θέλαμε και εμείς τις δικές μας προτάσεις για ποσά να ψηφιστούν. Δεν είμαι σίγουροι για τη σειρά που πρέπει να ψηφιστούν, αλλά θέλουμε οι παρατηρήσεις, τα σχόλια ξεχωριστά να ψηφιστούν. Λοιπόν, η συντονία έχει το λόγο. Τώρα βλέπω ότι έχουμε ένα, μια τροπολογία για να σβήσουμε τη γραμμή, οπότε αυτή θα πρέπει ε, η 829 να ψηφιστεί πρώτα. Άρα, καταρχήν ε, βάζουμε την πιο επαχθή ε, τροπολογία πρώτα την 629. Ε, ε, ποιος είναι υπέρ. Πέντε είναι οι κακοί. Ποιοι... Έξι, έξι. Ποιοι είναι ε, κατά. Αποχές. Άρα απορρίπτεται αυτή η τροπολογία, οπότε έχουμε να ψηφίσουμε την 628 που είναι κάπως λιγότερο κακιά. δηλαδή το απόγευμα, η συγκήτρια. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ψηφίσουμε την 829 ε, γιατί αυτή είναι η πιο γενναιόδορη. Και εγώ είμαι κατά. Αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, η τροπολογία 829 ε, πρώτα είναι ο αριθμός που απέχει περισσότερο από τη θέση του εισηγήτρες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Οι περισσότεροι είναι κατά, διότι δεν ακολούθησαν τη θέση των σοσιαλιστών άλλοι, άρα απορρίπτεται η 829. Οπότε, το 482. Συμφωνείτε. Ποιος είναι για το 482. Κατά. Αποχές υπάρχει μια πλειοψηφία υπέρ του 482 οπότε επικαλύπτει τις δύο επόμενες τροπολογίες αλλά πρέπει να επανέλθουμε στην 628 εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα αλλά αφού εσείς καταλαβαίνετε σας ακολουθώ 628 λοιπόν μόνο παρατηρήσεις και τι μας λέει ο εισηγητή, εισηγήτρια σχετικά δεν θέλει και ο, ο, ο Κέσαρα ζητά θαλάτωση ε, του νο, μονομάχου. Ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν για το 628. Και, και το ΕΛΚ δεν ακολουθεί την εισηγήτρια. Ψηφίστε λοιπόν. 21 υπέρ, 13 κατά, 2 ε, αποχές, άρα οι παρατηρήσεις αυτές εγκρίνονται. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχουμε καλύψει όλη αυτή την γραμμή για το EGF, για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Το 31-30 καλύπτεται και το 4705 η υπόλοιπη σελίδα είναι ο συνήθις Χάουζερ δηλαδή απορρίπτεται είμαστε τώρα στο 28 το οποίο η ε, σελίδα 28 η οποία καλύπτεται ολόκληρη αντιθέτως στη σελίδα 29 το 152 για τους οργανισμούς δεν καλύπτεται και πρέπει να το ψηφίσουμε η εισηγήτρια είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ. Δύο υπέρ. Κατά. Πολύ. Αποχές. Απορρίπτεται. Η υπόλοιπη σελίδα καλύπτεται από τις τροπολογίες μας για τους οργανισμούς, επίσης το European Maritime Safety Agency, αλλά όσον αφορά την αηφόρο ανάπτυξη πρέπει να ψηφίσουμε το 394. Ε, η συγγήτρια είναι κατά. 394 ποιος είναι υπέρ. Η πράσινη. Κατά. Πολύ. Άρα απορρίπτεται. Αλλά η συγγήτρια είναι υπέρ της 155 για αυτό το οργανισμό. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές το 155 λοιπόν υιοθετείται μου λέγουν ότι συνδέεται με το 156 393 πρώτα για τα μέτρα εναντίον της ρήπανσης. Η συγγήτρια κατά υπέρ είναι η πράσινη. Κατά αποχές. Άρα οι περισσότεροι θέλουν τη ρήπανση και απορρίπτουν την τροπολογία 394. Το, ε, το, ε, το 156 ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στο <clears throat> κεφάλαιο 03. Η τροπολογία 157. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 157 στο κάτω μέρος της σελίδας 30. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μαρκοπόλο 2. Μου λέγουν ότι πλέον δεν μπορώ να ψηφίζω. 41-39 τροπολογία. Απερίφη το 158 της Επιτροπής Μεταφορών, η συγγήτρια είναι υπέρ, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Μία, α, κατά μία αποχή εγκρίνεται. Η ολοκλήρωση του προγράμματος Μαρκοπόλο 41-40. Είναι μια κατα μια αποχη τροπολογία του κυρίου Χάρτον, άρα Χάρτονγκ, αρα απορριπτεται το, η υπόλοιπη σελίδα καλύπτηκε από την τροπολογία για τους οργανισμούς. Γυρίζουμε σελίδα, σελίδα 32, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε την 159, η συγγήτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Μία υπέρ, όλοι οι άλλοι κατά. Άρα απορρίπτεται. Η ασφάλεια των μεταφορών 160. Η συγγήτρια είναι υπέρ της 160. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Οι μεταφορές θα είναι ασφαλείς. Ε, στο τέλος της σελίδας έχουμε τα πιλωτικά προγράμματα. Περνάμε στη σελίδα 33 και στην αρχή έχουμε την τροπολογία 622 τούνελ μεταξύ Σουηδίας και Δανίας ο εισηγητής δεν είναι υπέρ αυτής, αυτού του τούνελ. Ποιος είναι υπέρ? 622. Οι Δανέζοι είναι υπέρ, οι Σουηδές είναι κατά. Θα κάνουν δηλαδή το μισό τούνελ. Λοιπόν, 622. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ο Γκέραν λοιπόν ακολουθεί την πειθαρχία, δεν ε, χρηματοδοτεί το τούνελ, οπότε καταπίπτει το 43-47, αλλά η 161. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρα οι επόμενες δύο καλύπτονται. Το Σεζάρ 162. Άβε Σέζαρ. Ποιο είναι υπέρ του Σέζαρ. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιο είναι κατά. Ο, ο Βρούτος σήκωσε χέρι. Λοιπόν, ο, Σεζάρ, ο Κέσαρας, το Σεζάρ δηλαδή, επεβίωσε ε, μεταφορές ε, ε, και έρευνα 163. Ποιος είναι υπέρ, κατά εγκρίνεται. Και μπορώ πάλι να ψηφίζω και ξαναβρίσκουμε το Σεζάρ με την τροπολογία Χάρτονγκ που απερίφθη 164 υπέρ της Σεζάρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Το 164 εγκρίνεται. Γυρίζουμε σελίδα. Και στην αρχή έχουμε στο European Research Council Executive Agency και στη Research Executive Agency όλα αυτά καλύπτονται αλλά στη γραμμή Expenditure Related to Research Staff πρέπει να ψηφίσουμε 41-43 τροπολογία του χάρτων που απορρίπτεται ο συνήθως 510 ε, υποβάλλουμε προς ψήφιση η συγκήτρια είναι κατά ποιος είναι υπέρ κατά Πολλοί άλλοι. Λοιπόν, απορρίπτεται. 46-23 Χάουζερ είναι συνηθισμένη. Άρα δεν την ψηφίζουμε, απορρίπτεται. Περνάμε σελίδα 35. Πρώτη τροπολογία Χάρτονγκ απορρίπτεται και ψηφίζουμε την 82 που εγκρίνει η συγγήτρια. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και καλύπτει την τροπολογία Σούριαν. 504 καινοτόμα ιατρική. Η συγγήτρια είναι κατά της καινοτόμας ιατρικής. Ποιος είναι υπέρ. Κατά όλοι αποχές οπότε δεν θα έχουμε καινοτόμα ιατρική 41-43 χάρτον απορρίπτεται συνήθως 83 83 η συγγήτρια είναι υπέρ ποιος είναι υπέρ κατά μία ψήφος δύο, κατά εγκρίνεται 42-84 καταπίπτει 42-44 είναι πιλωτική δράση άρα δεν την ψηφίζουμε και είμαστε στη σελίδα 36 πίσω συνήθις τροπολογία Χάρτονγκ απορρίπτεται τροπολογία 503 ο Ισεγίτρα είναι κατά ποιος νιπέρ. μία ψήφος κατά αποχές απορρίπτεται 421 Καταρχήν οι αριθμοί. Οι συγγήτροι είναι υπέρ των αριθμών. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Τρεις. Αποχές. Άρα οι αριθμοί του 421 εγκρίνονται. Όσον αφορά τα σχόλια, η συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Η φιλελεύθερη. Αποχές το βάθος της εθούσης οπότε πάλι τα α, σχόλια υπερψηφίζονται με διαφορετική πλειοψηφία. Και τώρα περνάμε στις νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες που χρειάζονται ε, μέγα χρηματοδότηση. Nanoscience για μέγα ε, χρηματοδότηση. Ποιος είναι υπέρ, η συγκήτρια είναι υπέρ. Κατά. Τρεις κατά, αποχές, 85 υιοθετείται, 133. Πιλωτική δεν τη συζητάμε και φτάνουμε Cooperation Energy, 587. Δεν τη θέλει η συγκήτρια. Ποιος είναι υπέρ. Χωριστή ψηφοφορία. Τι θεωρεί η συγκήτρια για τους αριθμούς δεν της αρέσουν. Ποιος είναι υπέρ. Κανείς. Μάλλον η πράσινη. Οι δύο πράσινοι. Ο ένας κύριος, μία κυρία. Ποιος είναι κατά. Όλοι οι υπόλοιποι δυστυχώς. Αποχές, Αλλά πάνε οι αριθμοί. Αλλά υπάρχουν και σχόλια. Ποιος είναι υπέρ των σχολείων. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα σχόλια του 600, 587 μπορώ ή δεν μπορώ να ψηφίσω. Ο Ζων Λίκ έφυγε, άρα εγώ μπορώ να ψηφίσω. Όλοι ψήφισαν, τέσσερις κοιμούνται ακόμη. 23 κατά, 14 υπέρ, άρα απορρίπτεται. Χωρίς σχόλια λοιπόν. Είναι μια τροπολογία χωρίς ούτε αριθμούς, ούτε σχόλια, άρα δεν υπήρξε ποτέ. 87, μόνο αριθμοί. Η συγκίτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κανείς δεν το θέλει. Όλοι κατά, άρα διαγράφεται. Το 86. Εδώ η συγκίτρια είναι υπέρ, δεν την διαχωρίζουμε και την ψηφίζουμε όλοι μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ξαναγυρίζει ο Ζων Ντεν. Μπορώ να συνεχίσω να ψηφίζω, ωραία. Η 4282 καλύπτεται, η 428 include bio-coal production from wood waste. Αρέσει στην εισηγήτρια που είναι υπέρ. Τι ποιος είναι υπέρ. Το ΕΛΚ ε, δεν υπάρχει πια. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην επόμενη γραμμή. Fuel cells and hydrogen joint undertaking. Εισηγείται υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 89. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία κόμιλάδα. Για τα πιλωτικά θα τα ξαναδούμε. Και είμαστε σελίδα 38. Ε, cooperation in environment including climate change. Έχουμε τη συνήθη τροπολογία χάρτων που απορρίπτεται. 717 εισηγείται είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Άρα πρέπει να προβούμε σε ηλεκτρονική ψηφοφορία και έχω δικαίωμα να ψηφίσω. Ψήφισαν 39 από 42, άλλοι κοιμούνται. 25 κατά, 14 υπέρ. Άρα απορρίπτεται. 42-81. Η συγκήτρια υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται και καλύπτει το 90. Επόμενη γάμη 91. Ε, η συγκίτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συνεργασία ε, Cooperation ε, in Transport Including Aeronautics υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρα καλύπτει και την επόμενη προς μεγάλη χαρά του Λάσλο Σούριαν. Περνάμε στην 93. Η συγητή είναι υπέρ για να έχουμε καθαρό αέρα. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά. Τρεις. Ποιοι απέχουν, άρα εγκρίνεται η 93 και καλύπτει και την επόμενη και ξαναβρίσκουμε τα fuel cells and hydrogen που παρισφρίουν παντού με την 507 που δεν αρέσει στον εισηγητή ποιος είναι υπέρ. Τέσσερις. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Απορρίπτεται. 94. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συνεργασία στις κοινοοικονομικές και ανθρώπινες επιστήμες. Η 41-43 είναι του κυρίου Χάρτον απορρίπτεται. Η 500 δεν αρέσει στην εισηγήτρια. Ποιος είναι υπέρ. Τέσσερις. Κατά. Πολύ. Άρα απερίπτεται η 595. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και καταλήπτει την 4278. Για την 631 πρέπει να υποβάλουμε στην ψηφοφορία τα σχόλια. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Η συγγήτρια είναι υπέρ αποχές εγκρίνονται τα σχόλια και η 4368 ήταν ταυτόσιμη και περνάμε στο Rix Sharing Finance Facility που ικανοποιεί την εισηγήτρια 96. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρα καλύπτει και την επόμενη και περνάμε στην επόμενη σελίδα 40 στο, στον απίθανο τίτλο «Ideas», ιδέες. 41-43, συνήθως τοπολογία χάρτων απορρίπτεται και για να χρηματοδοτηθούν οι ιδέες προτείνει η συγγήτρια την 97. Ποιος είναι υπέρ των ιδεών. Κατά αποχές εγκρίνεται και καλύπτει τις δύο επόμενες τροπολογίες. Περνάμε στο Capacity Research Infrastructures 718. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές ε, εξαφανίζεται. Αλλά για την 98 η εισηγήτρια είναι υπέρ. Ποιος άλλος είναι υπέρ με την εισηγήτρια. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και καλύπτει την επόμενη. Στη συνέχεια υπάρχουν πιλωτικά σχέδια, δεν τα συζητάμε, πάμε 41. Capacity Research for the Benefit of Small and Medium Size Enterprises. Έχουμε πάλι τροπολογία Χαρτών 41-43 που απορρίπτεται, 719 που δεν αρέσει στον εισηγητή, ποιος είναι υπέρ. Κανείς. κατά, άρα διαγράφεται. Η 543 αντιθέτως έχει τη στήριξη της συγκήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και καλύπτει τις επόμενες δύο. Περνάμε στην επόμενη γραμμή. Τροπολογία 100. Αρέσει τον εισηγητή ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καλύπτει και την επόμενη 41-43 Capacity Research Potential απορρίπτεται. 101 της Επιτροπής Βιομηχανίας. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καλύπτει και την επόμενη. Επόμενη, Science in Society. αρέσουν οι εισηγητή. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται και καλύπτει και την 4271. International Cooperation Activity 103 εισηγήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και καλύπτει και την επόμενη ξαναβρίσκουμε την Risk Sharing Finance Facility 104. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και καλύπτει την επόμενη. Περνάμε εις την ε, γραμμή Support for Coherent Development of Research Policies. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και καλύπτει και την 4268. Ερα ευρατών 587 των ε, πρασίνων που δεν είναι για τη σύνδεξη. Κατά. Η πράσινη υπέρ και όλοι οι υπόλοιποι κατά. Άρα η τροπολογία απορρίπτεται. Η 587 ψηφιστεί τώρα ή αργότερα. Εισηγήτρια, θέλετε να ψηφίσουμε αυτήν την τροπολογία για την ΙΤΕΡ. Είμαι πεισμένη ότι θα έπρεπε να θέσουμε σε ψήφιση την τροπολογία όπως έχει κατατεθεί από τους πράσινους. Είμαι κατά αυτής της τροπολογίας, αλλά θα πρέπει να την ψηφίσουμε. Άλλα λόγια. Αν κατάλαβα την πολιτική σκοπιμότητα, η συγγήτρια θέλει να χρησιμοποιήσει την γραμμή ΙΤΕΡ για να χρηματοδοτήσει άλλες προτεραιότητες. Πράγμα το οποίο προϋποθέτει ότι πρέπει να κρατήσουμε τα χρήματα που είναι στη γραμμή ίτερ. Ενώ η τροπολογία 587 των Πρασίνων διαγράφει αυτό το ποσό και την δυνατότητα για τον εισηγητή να το χρησιμοποιήσει αλλού. Γι' αυτό και ο εισηγητής θέλει να διατηρήσει αυτή τη χρηματοδότηση και προτείνει να θέσουμε προς ψηφοφορία την 587 και να την καταψηφίσουμε. Καλά κατάλαβα αυτό είναι ο χειρισμός που θέλετε να κάνετε. Ζητάτε το λόγο. Κυρία Εισηγήτρια. Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπατε. Πρέπει επίσης να επανέλθω σε αυτό που πόσο κομψά το αποκαλέσατε. Αυτό το καγέ, αυτό το τετράδιο, το φυλάδιο για το έγγραφο, για το στη σελίδα 12 έχω καταθέσει την 3.000 τροπολογία ως εισηγήτρια. Είναι μια τροπολογία που μπορούμε να την ψηφίσουμε α, αύριο, όπως είπα πιο πριν. Έχει κατατεθεί για την μείωση του ΙΤΕΡ κατά 45 εκατομμύρια ευρώ και προφορικά μπορεί να προσαρμοστεί αν χρειαστεί όταν θα ψηφίσουμε αύριο. Αυτά όπως είπατε αύριο. Ο κύριος Έλλης θέλει το λόγο. Είναι μόνο για αυτό το θέμα του Ήτερ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι λαμβάνουμε αποφάσεις χωρίς να ξέρουμε υποχρεωτικά το συνολικό πλαίσιο αυτής της απόφασης για την χρηματοδότηση και τις υποχρεώσεις που έχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση για διεθνή όργανα, διεθνή θεσμικά όργανα όπως η ΙΤΕΡ. Ευγνώμων θα, ήθελα, θα ήμουν αν ήξερα ποιε είναι οι δεσμεύσει για πληρωμές ώστε να έχουμε μια βάση για συζήτηση αύριο, να ξέρουμε τι κάνουμε. Ευχαριστώ. Oui, merci, James. Ε, Ευχαριστώ δεν ήσασταν εδώ, αλλά χθε το βράδυ κάναμε μία εκτενή συζήτηση για το ΙΤΕΡ. Συνοψίζω το συμπέρασμα των εισηγητών και συντονιστών λέγοντας ότι πάει μία αρκετά ευρία στήριξη, όχι ομοφωνία γιατί ορισμένοι είναι ενάντι για να στηριχθεί αυτή η πρωτοβουλία. Επίσης, ε, η κατάσταση στο Συμβούλιο είναι πολύ συγκεχημένη όσον αφορά τις ε, ε, επιπρόσθετες ανάγκες του ΙΤΕΡ και πότε θα χρειαστούν άλλες πιστώσεις. Οπότε, στα πλαίσια μιας πολιτικής τοποθέτησης που επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να διαπραγματευτεί με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, Υπάρχει μία συμφωνία των εντολοδόχων για να μας να συμφωνήσουμε επί τη στρατηγική που προτείνει η συντονία και ε, θα αποφασίσουμε αύριο για το ποσό. Άρα το 587 ε, ποιος είναι υπέρ, η συγκήτρια είναι κατά. Η πράσινη και η κυρία Ανδρέασεν. Ποιοι είναι κατά? Όλοι οι υπόλοιποι. Αποχές. Άρα η 587 απορρίπτεται. 584 ε, στην ε, σχάση, πυρνική σχάση. Η συγγήτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. ακόμη και για τους πράσινους δηλαδή δεν υποστηρίζουν την τροπολογία τους, την υποστηρίζουν. Κατά εγκρίνεται. Όχι, όχι, όχι, με συγχωρείτε, απερίφθη. Ε, εγώ είμαι ε, θύμα των ακτινοβολιών. Ε, τώρα, η επόμενη είναι κλασική Ερενχάουζερ και οι δύο επόμενες στη σελίδα και γυρίζουμε σελίδα. Είμαστε σελίδα 44, έχουμε τη 41-44 τον κυρίο Αχάρτον που απορρίπτεται. Το ίδιο ισχύει και για την 47-66, όχι. Ψηφίζουμε τη 47-66 Χάουζερ, που είναι αντίθετη, η συγγήτρια είναι κατά. Ποιος είναι κατά, απορρίπτεται. Επόμενη γραμμή. Τροπολογία Χάρτογκ, η οποία θεωρείται ότι απερίφθη, 106 συγγήτρια είναι υπέρ, ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ της 106, ποιος είναι κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Επόμενη γραμμή, 41-44 χάρτων θεωρείται ότι απερίφθη, 46-27 Χάουζερ απορρίπτεται, συνήθις, 131. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Safer Internet Program γραμμή. Συνήθι τροπολογία χάρτων απορρίπτεται 4362 από τον Αντιπρόεδρο Αλβάρο. Στηρίζεται από την εισηγήτρια. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έπαψαν να ψηφίζουν οι πράσινοι. Γυρίζω σελίδα 45. Ερενχάουζεν 4663 διαφορετική για αποθεματοποίηση η εισηγήτρια είναι κατά. Κατά. Κανείς δεν το στηρίζει. 4659. Πρέπει επίση να ψηφίσει η εισηγήτρια κατά ποιος νιπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Επόμενη γραμμή. ICTSP. 41-44 συνήθις χαρτόγκ οπότε απορρίπτεται 697 ο εισηγητής είναι κατά ποιος νιπέρ. κατά αποχές ε, διαγράφεται 108 έρχεται από την Επιτροπή μας της Βιομηχανίας αλλά δεν αρέσει στην εισηγήτρια ποιος είναι υπέρ. Κανείς υπέρ διαγράφεται. 107. Αυτή αρέσει στην εισηγήτρια. Ποιος είναι υπέρ. 12. Ξυπνήστε. Κατά. Αποχές. 107 εγκρίνεται και καλύπτει την επόμενη αλλά όχι την 422. Οπότε θέτω προς ψήφιση την 422 μόνο τις παρατηρήσεις σχετικά με το 112. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και ο Σαλβαντόρο ε, ε, ευχαριστεί την Επιτροπή ε, Προπολογισμού. Στην επόμενη σελίδα το 4100 δεν ψηφίζεται. Το 41-44 συνήθις άρτων θεωρείται ότι απερίφθη. 109 ψηφίζουμε, η συγκίτρια είναι υπέρ, ποιος είναι υπέρ. χερ, Αποχές. Εγκρίνεται. Άρτο 42-66 καλύπτεται. Περνάμε στο πρόγραμμα Artemis, Artemis Joint Undertaking, μία στιγμή ποιησης. Τροπολογία 110, ε, η είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά της Artemis. Αποχές, η Artemis θα έχει και φαρέτρα και τόξα. Καλύπτει και το επόμενο. Και ξαναπερνάμε σε στήριξη του προγράμματος Άρτεμις. Ποιος είναι υπέρ του 111. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και καλύπτει και την επόμενη. Είναι Joint Undertaking 112 που προτείνει η συγγήτρια. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και καλύπτει και την επόμενη. Support expenditure for ENIAC joint undertaking 113 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και καλύπτει και την επόμενη. Και φτάνουμε στο capacity research infrastructure. 41-44 συνήθιση χάρτων να απορρίπτεται. 114 ψηφίζεται ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. και καλύπτει και την επόμενη γιατί και Στη συνέχεια έχουμε Χάρτονγκ Σαντέν 45 που θεωρώ ότι απερίφθηκε. και το ίδιο ισχύει και για την Έρεν Χάουζερ 47-65. Γυρίζω σελίδα. External Staff for Research. Πρώτη τροπολογία 41-45 του κυρίου Χάρτονγκ απορρίπτεται. Μετά τα επόμενη γραμμή 10.01.05.03 ε, ε, απορρίπτεται η τροπολογία χάρτων και έχουμε και μία τροπολογία συνήθη Ερενχάουζερ και άρα θεωρούμε ότι απορρίπτεται. Ε, μετά φτάνουμε στη γραμμή 10.02 Directly Finance Research ο Operation Appropriation, 819 τροπολογία της ΓΚΟΕ, αντίθετος συγητής, ποιος είναι υπέρ. Βλέπω ότι οι σοσιαλιστές είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Ε, αλλά οι υπόλοιποι είναι κατά, μόνο οι σοσιαλιστές έμειναν και δεν εγκρίνεται. Οι 834 είναι ίδια. Το σχόλιο είναι διαφορετικό. Αποκλεισμό ε, για την έρευνα για τους ε, Ισραηλινούς στρατιωτικούς. Η είναι κατά ποιος είναι Οι σοσιαλιστές. Κατά. Πολύ. Άρα απορρίπτεται. Δεν έχουμε δηλαδή καμία τροπολογία στην 10.02. 10.02.01. 41-45 συνήθει χάρτων που θεωρώ ότι απορρίπτεται. 115. Ο εισηγητή είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ. Εγκρίθηκε. Η επόμενη κατήπτεται. Σελίδα 49. 116 εισηγήτρια υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται επόμενη καλύπτεται. Θα ψηφίσουμε όμως τα σχόλια, remarks, τις 15.84 υπέρ. Οι πράσινες κατά, οι άλλοι αποχές, τα σχόλια απορρίπτονται τις 5.84. Έρνχαρ χάρος συνήθις απορρίπτεται. 35 η συγκέντρια υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ η συγκέντρια υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 πιλωτικό αργότερα όλη η επόμενη σελίδα η 50 αγγλική καλύπτεται από τις υπηρεσίες και 51 52. Καλύπτεται από τις υπηρεσίες. Στο κάτω μέρος της 53. Implementation and Development of the Internal Market. Σε 683 καλύπτεται. Ή σε 684 καλύπτεται. Η 38. Σε 683 συνήθισε Ερενχάουζερ απορρίπτεται. 39 ψηφίζεται. Η 39. Υπέρ. Η υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 549. Τελωνία 2013. Αποσύρεται. Δεν θα έχουμε τελωνία το 2013. Φυσκάρις 2013-326. Η συγκεκριά δεν της αρέσει. Ποιον του αρέσει το φυσκάρις. Η πράσινη. Ούτε, ούτε καν η πράσινη. Α, ναι είναι. Ο κύριος Αλφονσίν είναι υπέρ. Κατά Όλο ο κόσμο Και η κυρία Τρίπελ. Η πράσινη είναι διαρριμένη στο φρατό φυσικά τη. Απορρίπτεται. 2.65 καλύπτεται. Το πρώτο μέρος της σελίδα 54 καλύπτεται μέχρι το European Institute of Innovation and Technology Structure. Μιλάω για την 117, εισηγήτρια υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η επόμενη καλύπτεται lifelong learning καλύπτεται με εξαίρεση την 312 Υπάρχει μια παρατήρηση. Τα σχόλια, τα σχόλια. Η συγκίτρια είναι υπέρ του σχολείου. Πώς είστε υπέρ του σχολείου. Κατά. Κάμποση. Αποχές. Πλειοψηφία υπέρ. Εγκρίνεται το σχόλιο του Προέδρου Κάρλο Καζίνη. Το υπόλοιπο είτε καλύπτεται είτε πιλωτικά. Αύριο αυτά. Σελίδα 56. Στο κάτω μέρος της σελίδας ένα Έρεν Χάζερ που πρέπει να ψηφίσουμε γιατί είναι ασύνηθες να μπει στο αποθηματικό. 46-48 υπέρ. Κανένας δεν είναι υπέρ. Α, μόνο ένας μόνο. Κατά όλος ο κόσμος αποχές απορρίπτεται. πιλωτικά μέχρι η γραμμή που έχει το εξαιρετικό ε, τίτλο People, People. Εδώ έχουμε τις 41-48 χάρτων, συνήθις απορρίπτεται. Και υπέρ των People έχουμε το People's Party, το οποίο είναι λογικό, 540. Η υπέρ, κατά του People's Party, ευχαριστώ, αποχές, εγκρίνεται και καλύπτει την τροπολογία Αμπανταμιέν. 3.15 ψηφίζουμε. Μόνο τα σχόλια. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκαν τα σχόλια. Το υπόλοιπο καλύπτεται. Σελίδα 58 πολύ ωραία σελίδα διότι δεν μας ενδιαφέρει. Τα μισά είναι πυροτικά προγράμματα και τα άλλα μισά καλύπτουν τις υπηρεσίες. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για το μεγαλύτερο κομμάτι της 59. Ξαφνικά όμως εμφανίζεται μια τροπολογία 328 που πρέπει να ψηφίσουμε. Εισηγήτρια υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Τα υπόλοιπα δεν μας ενδιαφέρουν. Αργότερα αυτά. Σελίδα 60 πάνω. Broadband Internet in Rural Areas. Θα θυμόστε είναι το πρόγραμμα ανάκαμψης. Έχουμε η τροπολογία 132 για νέα γραμμή. Συγήτρια είναι κατά υπέρ. Κανένας. Κυρία Βέρτμαν μόνο. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4608 Ερενχάουσερ κλασική. Απορρίπτεται. Για το MIDS καλύπτεται. EU Statistical Program χάρτουμ συνήθες απορρίπτεται. Το υπόλοιπο καλύπτεται. Το ίδιο και η αρχή της 61. «47-15 είναι χάζερ λίγο διαφορετική, την ψηφίζουμε. Όχι, αυτό είναι στο 10% απορρίπτεται. 47-16 το ίδιο. Το υπόλοιπο καλύπτεται. Πάει 61. Σελίδα 62. Η πρώτη καλύπτεται. Η δεύτερη ένα κλασικη κλασική απορρίπτεται. 41-50 Χάρτον κλασική απορρίπτεται. 44-93 Έιντερ Γκαρθία Θάμπαλ. Καρδιά Θάμπαλ. Ψηφίζουμε. Η δεν της αρέσει. Υπέρ. Αϊάν θέλει το λόγο. Χωριστή ψηφοφορία. Χωριστά το νούμερο, το ποσό, χωριστά τα σχόλια. Ωραία, πρώτο το ποσό. Της 4493. Η συγκίτρια τι μας λέει. Κατά. Ποιος είναι υπέρ Το ποσού. Κατά αποχές Μόνοι οι είναι υπέρ τα σχόλια τώρα η κατά υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ για τα σχόλια απορρίπτεται με 23-16. Αυτή η τροπολογία δεν έχει ούτε ποσό, ούτε σχόλια. Τι να κάνουμε. 123 συγγύτρια υπέρ. Υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίθηκε. 140. Creation of a supergrid. Η Εξακολουθώ να βρίσκομαι σε κατάσταση ματέωσης γιατί δεν μπορώ να ψηφίσω. Ψηφίζουμε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, παργά όμως, παρακαλώ πιο γρήγορα. Ψηφίστε. Άντε μια προσπάθεια ακόμα. Μαστίγιο δεν έχω. Πέρας. 20-20. Απορρίβεται. Αν μου είχατε επιτρέψει να ψηφίσω κι εγώ, δεν ξέρω τι θα, αποτέλεσμα θα είχαμε. Προειδοποιώ τους τεχνικούς τα αποτελέσματα της ψήφου. Εγώ τα έχω, αλλά οι άλλοι δεν τα έχουν. Κάνουμε μια εικονική ψηφοφορία, παρακαλώ, μια εικονική ψηφοφορία. Ποιο είναι υπέρ. Υπέρ της εισηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ της εισηγήτριας. Εγώ ψηφίζω. Ψηφίστε όλοι. Είμαστε 43 παρόντες και μόνο 36 ψηφίζουν. Τεμπέλιδες είστε. Πέρας. Πάλι δεν βλέπετε. Τι όλες στημένες, στημένες ήταν όλες τις ψηφοφορίες, θα τις ξανακάνουμε. Ωραία γίνεται. Τι σας φτιάχνει. Που τώρα ξέχασε πού ήμασταν. Support activities. 124. στο κάτω μέρος της σελίδα 62 αγγλικά. Συγήτρια υπέρ υπέρ. Κατά. άποχε Εγκρίνεται. Μετά έχουμε την 63. Θα το ψηφίσουμε όλα εδώ. 134. Τα δύο 134 στην αρχή, European Wind Initiative και European Solar European Initiative, δύο διαφορετικές ψήφους. Μία καταρχήν για να γίνει γραμμή και μία για το ποσό. Μπορούμε να ψηφίσουμε και τα δύο ταυτόχρονα, και όποιος είναι υπέρ του, της αιωλικής είναι και υπέρ του ήλιου. Λοιπόν, για την σύσταση των γραμμών. Οι δύο τροπολογίες μαζί, 134 Γητρα είναι κατά η ηλεκτρονικής ψήφος και τώρα θα δείτε και το αποτέλεσμα αυτή τη φορά. Ένας παραπανήσιος στο ΕΛΚ. Δεκαοχτώ-δεκαεφτά απορρίπτεται. Το ΕΛΚ είναι κατά. Δεν είναι στημένο το αποτέλεσμα, το βλέπετε στον πίνακα, συμφωνείτε. Η αρχή της γραμμής αυτών των δύο γραμμών εγκρίνεται καταρχήν και για την άνεμο και για τον ήλιο. Τώρα το θέμα είναι τι νούμερο βάζουμε. Βέβαια που είναι κατά της γραμμής πιστεύω είναι η ίδια πλειοψηφία. Θα ξαναψηφίσουμε. Αυτή τη φορά θα αφαιρέσουμε έναν του ΕΛΚ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τώρα ούτε δεν δέχνουμε. Ε, θα κάνουμε τη γραμμή χωρίς ποσό. Ούτε άνεμος, ούτε ήλιος. Υπάρχει γραμμή. Μια μέρα όταν θα έχουμε άνεμο ή ήλιο, τότε βλέπουμε. Πολιτικά είναι ε, ε, υποστηρίξιμη αυτή η θέση. Τώρα, Μπορούμε με το ίδιο έτσι κλίμα να ψηφίσουμε, έχουμε το άνεμο, να ψηφίσουμε unblock όλη την υπόλοιπη σελίδα. Τι λέτε. Όλα τα 134 μέχρι κάτω. Τι λέτε. James. Μια από τις γραμμές είναι η European Solar European Initiative. Την κάναμε τη γραμμή χωρίς ποσό. Θα μπορούσαμε να τη βάλουμε προ memoir. Ξέρω, στο μέλλον ενδεχομένως θα μπορούσαμε να το χρηματοδοτήσουμε. Πρόεδρος, με αυτός είναι ο στόχος αυτής της τροπολογίας. Ο άνεμος μας τελείωσε. Ψηφίσαμε. Έλλης, κύριε Πρόεδρε, έχουμε δύο γραμμές εδώ. European Solar Initiative δύο φορές. 134. Προτείνω να το βάλουμε προμέμορα. Ψηφίσαμε να μην πει ποσό. Δεν είναι σαφές αυτό. είναι διαφορετικά. Ψηφίσαμε τις δύο πρώτες γραμμές. Ένα pour mémoire, χωρίς νούμερο, χωρίς ποσό, για τον άνεμο. Τώρα ψηφίζουμε en bloc τις τέσσερις τροπολογίες, τις τελευταίες. Γραμμή mémoire, υπέρ. Ή ηλεκτρονικά. Ψηφίστε μας λείπουν λοιπόν, κόσμος. Μερικοί δεν θέλουν να ψηφίσουν. 40, 41. Ένας ΕΛΚ παραπάνω. Έφυγε το ένας του ΕΛΚ. Ωραία. 20 υπέρ, 18 κατά. Εγκρίθηκαν αυτές τις τροπολογίες. Γυρίζω σελίδα. 64. Η αντιπρόεδρος προσπαθεί να περισπάσει την προσοχή του Έλκ από την πλάτη μου. Σελίδα 64. Ένα πρόγραμμα για το Intelligent Energy. Υπάρχουν και αυτά. Το έχουμε συναντήσει. Υπάρχουν. 41-50 χάρτον κλασική απορρίπτεται 7-20 εισηγήτρια κατά υπέρ κατά ευχαριστώ αποχές απορρίπτεται 126 εισηγήτρια υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η επόμενη καλύπτεται 125 Συγγήτρια υπέρ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η επόμενη καλύπτεται. 582. Νέα γραμμή. Προμεμόρια. Η συγγήτρια δεν το θέλει. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 582. 39, 40, stop. 24 16 υπέρ απορρίπτεται. 127 εισηγήτρια υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προπολογία της ε, Χριστίνα πιλωτικό η επόμενη σελίδα, 136. Nuclear safety. Decommissioning. Τι λέει η συγγετριά. Πρέπει να ψηφίσουμε. Όπως είναι η σειρά πρώτη, 651 αν εγκριθεί η 128 καταπίτη. Τι είστε, είστε υπέρ ή κατά. Όχι, είμαι υπέρ του 651. 6.51. πενήντα ένα. Η συγκέντρια είναι υπέρ, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 128 καταπίπτει. Έρευνα σε σχέση με την ενέργεια. 41-50 συνήθις χάρτογα. Απορρίπτεται. 130. Συγκίτρια υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οι τρεις επόμενες καλύπτονται, αλλά όχι η παρατήρηση του 586 των πρασίνων. Η συγκέντρια είναι κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία 586. Τα σχόλια. Πέρασε. Απορρίπτεται με 27 επόμενη σελίδα. 41-50. Χάτον κλασική. Απορρίπτεται. 129. Εισηγήτρια υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η επόμενη καλύπτεται. Λοιπόν, το 2-1 τελείωσε και έτσι μπορούμε να εκδηλώσουμε τη συγκίνησή μας, την ικανοποίησή μας, υπό επιφύλαξη βέβαια, διότι πρέπει να δούμε, θα προσθέσουμε το τι ψηφίσαμε, τι συμπεράσματα θα μπορέσουμε να αποκομίσουμε αύριο για το σύνολο της γραμμής που αναφέρεται στο πρόγραμμα ITER. Και επιπλέον πρέπει να δούμε τα πιλωτικά προγράμματα. Κυρία εισηγήτρια, μπορούμε να περάσουμε τώρα στο 1β. Δηλαδή συμφωνούν οι εισηγητές να περάσουμε στο 1β. Μήπως ορισμένοι θέλουν να πλύνουν τα χέρια τους. Έχουμε χρόνο. Όχι. Δεν, δεν πλένουμε χέρια. θα πρέπει να κάνουμε όπως στο Αγγλικό Κοινοβούλιο. Αν κάποιος από το ΕΛΚ θέλει να πλύνει τα χέρια του, παίρνει και ένα σοσιαλιστή μαζί για να υπάρχει πολιτική ισορροπία. Λοιπόν, ερχόμαστε στο κεφάλαιο 1β, στην επικεφαλίδα 1β. Είσαστε όλοι έτοιμοι. Είμαστε στη σελίδα 66 ε, στο κάτω μέρος. Τροπολογία 384. Καλύπτεται για τους αριθμούς, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε τα σχόλια. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται τα σχόλια και ε, καλύπτουν και την επόμενη τροπολογία. Περνάμε σελίδα 67, η τροπολογία 469, η συγκήτρια υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καλύπτει τις δύο επόμενες. Στη γραμμή 040217, κλασική χάρτον που θεωρώ ότι απορρίπτεται η 821 της Γκουε. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έχουμε δύο τροπολογίες διαφορετικές. Του κυρίου Μπέλντερ, 4206, Εισηγήτρια. κατά, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ο κύριος Μπέλτερ έχει άλλη μία, ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Στο κάτω μέρος της σελίδας έχουμε την Χάρτονγκ που δεν είναι συνήθις, οπότε τη θέτω προς ψήφιση 41-30, η κίτρινη είναι κατά. Ο κύριος Χάρτον είναι υπέρ, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Είμαστε πάντοτε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στην αρχή της σελίδα 68, η 4131 συνηθισμένη χάρτον απορρίπτεται, 822 της ΓΚΟΕ εισηγήτρια κατά ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Βέβαια η ΓΚΟΕ αυτή τη στιγμή δεν εκπροσωπείται στις ψηφοφορίες. 449. Η συγγήτρια είναι κατά. Από το κανείς δεν τη θέλει, άρα διαγράφεται. 172 συγγήτρια υπέρ, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 172 υιοθετείται. Οι τρεις επόμενες ε, καλύφθηκαν. 41-32 χάρτον ξυνήθης απορρίπτεται. και καλύπτονται οι επόμενοι εκτός ε, από ότι τα σχόλια της 384 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 384. Και η επόμενη 384 για το Ταμείο Συνοχής. Ποιο ε, είναι υπέρ, είναι η ίδια τροπολογία, ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, η ίδια πλειοψηφία. Περνάμε στο Περιφερειακό Ταμείο, τροπολογία 376 της συγκήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι δύο επόμενες καλύπτονται. Έχουμε την 41-47 συνήθι χάρτων απορρίπτεται. Το ίδιο ισχύει και για την ε, και για το πις 41-47 θεωρούμε ότι περίφθη και πάμε στην σελίδα 70 385 ο εισηγητής είναι υπέρ ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οι τρεις επόμενες λοιπόν καλύφθηκαν και μου λέγεται ότι η 4356 έχει αποσυρθεί. Ο κύριος Χάγκλουμ την απέσυρε. Η 4311 ε, καλύπτεται της ε, Μπαλτζάνη Φραντζέσκα. Και έχουμε μια πιλωτική που θα δούμε αργότερα στο κάτω μέρος σελίδες και ξεκινάμε τη σελίδα 71. Ε, European Territorial Cooperation. συνηθις χαρτων χάρτονγκη 41-47 απορρίπτεται, 382 πρόκειται για σχόλια και αριθμούς. Transborder Cycling Networks, δηλαδή ε, διασυνοριακό δίκτυο ποδηλασίας. Το 382, ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. Αλλά καλύπτεται και αυτοί και οι δύο επόμενες. Καλά υπάρχουν άλλα σχόλια για την Macro Regional Cooperation, τη διατηρεί ο κύριος Χάρτογκ και ε, ο εισηγητής είναι υπέρ κατά αποχές η 4354 εγκρίνεται. Περνάμε στην επόμενη γραμμή. 391 Λογκέραν πριν. Σε αυτό το κονδύλιο για την τεχνική συνδρομή για το Περιφερειακό Ταμείο ανάπτυξη, έχουμε μια τροπολογία που είναι στην 13.03.43 λίγο υστερότερα τεχνική σύνδρομη και διάχυση πληροφοριών για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βαλτική θάλασσα. Το συζητήσαμε και θα προτιμούσαμε αν είναι δυνατόν αντί να δημιουργηθεί ένα νέο κονδύλιο να μεταφέρουμε τις παρατηρήσεις και αυτό που λένε για το τι θα έπρεπε να δοθεί στην, Βαλτική, στην περιοχή της Βαλτικής θάλασσας μέσω αυτής της γραμμής 0320 που είναι καλύτερη λύση από το να δημιουργηθεί ένα νέο κονδύλιο γιατί διαφορά θα έχουμε μια τεχνική συνδρομή για κάθε μακροπεριφέρεια που δεν είναι καλή ιδέα. Προτιμούμε αν είναι δυνατόν να έχουμε την τροπολογία 389 που θα εγκριθεί αλλά για την 130320. Ευχαριστώ. Madame είναι υπέρ. Ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο. Κατανοώ το σημείο, αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτήν την πρόταση. Ε, θα ψηφίσουμε όσο έχει, λέει ο κύριος ε, Χέρμαν. Ψηφίζουμε όπως είχε προβλεφθεί. 391. Η συγγήτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Η συγκίτρια είναι υπέρ. Άρα θα παραμείνει στη γραμμή αυτή. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Άρα εγκρίνεται η 391 και μένει εκεί που είναι. Ρυθμίσαμε το 583, όχι, πρέπει ε, να το καλύψουμε. One stop shop, αστείο ακούγεται υπάρχουν ε, υπέρ, οπότε ηλεκτρονική ψηφοφορία one stop one vote ε, κάνει λογοπαίγνιο ο πρόεδρος ο οποίος μπορεί να καταψηφίσει Λοιπόν, 21 υπέρ, 17 κατά, άρα ε, το One Stop ε, One Volt 583 καλύφθηκε, ε, το 4167 είναι πιλωτικό και μπορούμε να ανασάνουμε, η σελίδα 72-73 είναι πιλωτικά, εξαιρετικά. Και φτάνουμε τώρα στη γραμμή, ε, στην τροπολογία 389 που στηρίζει ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 373 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρα οι δύο επόμενες καλύπτονται. Cohesion Fund έχουμε το 505 που δεν αρέσει στον εισηγητή. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Macro Regional καινούριο το οποίο αποσύρεται. ...383 Cross Border Cooperation, πάλι διασυνοριακή ποδηλασία. Ποιο είναι υπέρ τη ποδηλασίας. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελειώσαμε με το 1β. Άρα ο κύριος Χάρτονγκ χειροκροτά. Κυρία εισηγήτρια, πιστεύετε ότι έχουμε οριμάσει, μπορούμε να πάμε στο 2, στο 3, να πάμε να φάμε, τι προτείνετε. Ουσιαστικά είμαι έτοιμη και πρόθυμη να ψηφίσουμε το τίτλο 2 Ανησυχώ όμως ότι ίσως δεν θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε μέχρι τη μία η ώρα αυτό το κεφάλαιο. Αν επιταχύνουμε όμως νομίζω μπορούμε να ψηφίσουμε τον τίτλο 2 και να τον καλύψουμε. On peut aller manger quand on parle d'agriculture. Bon. Bien. Ok, on profite du fait que Salvador n'est pas là pour décider qu'on commence heading 2. Tout le monde est prêt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 Ε, thank Φορική τροποποίηση για την τροπολογία 2.17. Σύστασή μου είναι να υπερψηφίσουμε, αλλά όχι για το ποσό που προτείνει η άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή, αλλά για το μισό 25 εκατομμύρια ευρώ και στο αποθεματικό όπω η πρόταση τη Άγκρη, αλλά το μισό των 25 να εγκρίνουμε ω κονδύλιο. Θέλετε λοιπόν απλώς να μειώσουμε στο ίμιση το απόθεμα, να κρατήσουμε τα 85 εκατομμύρια αλλά αποθεματοποίηση μόνο 25 τροπολογία του εισηγητή τροποποιήθηκε μένα, αλλά υπάρχουν ε, ε, συγκεχημένες ιδέες και κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Μπορώ να ψηφίσω ή όχι. Πρέπει να φτάσουμε τους 40. Ε, όχι. Κλείνει η ψηφοφορία. 16 υπέρ, 22 κατά, απορρίπτεται. Τους βλέπω τους πράσινους οι οποίοι χαίρονται. Ναι, ναι. Η γραμματεία μου λέγει ότι μπορούμε τότε να, εφόσον απορρίπτεται την προφορική ψηφοφορία, ε, τροπολογία να ψηφίσουμε τη γραπτή. Και επανέρχομαι στη 217 με τους αριθμούς. Κάποιος είναι υπέρ? Όχι. Απορρίπτεται, δεν το συζητάμε. Και τώρα είμαστε στο Intervention for Touch για το άμυλο, παρέμβαση για το άμυλο. Εγώ δεν ξέρω πέτνος πρόκειται, εσείς κάτι ξέρετε, υπάρχει μια τροπολογία χάρτων, οπότε καταψηφίζεται και διαγράφεται. Πάμε στην 575. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ της 575. Η πράσινη, κατά απορρίπτεται. Και πάλι έχουμε 575 πολλαπλή. Χρειάζεται να ψηφιστεί μια και καλή. Δηλαδή ε, απευθύνουμε στους πρασίνους, στη Χέλγα δέχεστε όταν ε, υπάρχει μία πολλαπλή τροπολογία 575 σε πολλές γραμμές μπορούμε να το ψηφίσουμε για όλες τις ε, γραμμές. Ωραία. Τότε ψηφίζουμε την 575 και θα εφαρμοστεί το αποτέλεσμα σε όλες τις επόμενες. Ποιος είναι υπέρ. Η πράσινη βέβαια. Και η Ιούτα. Και ο κύριος Χάρτον. Ποιος είναι κατά. Ε, άρα υπάρχει πλειοψηφία η οποία θα ισχύσει και αν υπάρξει ταυτόσιμη τροπολογία των πρασίνων. Και καλύπτει τις δύο επόμενες, μάλιστα, σε αυτή τη γραμμή. Και έρχομαι τώρα στη γραμμή Programs for Deprived Persons. Υπάρχει μία προφορική τροπολογία της εισηγήτριας. Η προφορική τροποποίηση είναι ως εξής. Στην τροπολογία 670 και λέει να ενταχθεί ένα ποσό 25 εκατομμυρίων ευρώ αντί 100 εκατομμυρίων. Και αυτό θα κάνει τις άλλες να καταπέσουν. Θα χαιρόμαστε αν μπορούσαμε να ψηφίσουμε ως έχει στον πίνακα ψηφοφορίας την απότερη τροπολογία πρώτα και μετά τις υπόλοιπες. So you could accept the rapporteur as a fallback. Θα μπορούσατε να δεχτείτε αυτό ως θέση αναδίπλωση ηγήτρια αν χάσετε την πρώτη ψηφοφορία, εντάξει. Σωστό. Donc, je soumets... Υποβάλλω λοιπόν Ε, ο εισηγήτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές. Η τροπολογία αυτή απορρίπτεται. Ο εισηγητής διατηρεί την πρότασή του, ναι. Ποιος είναι υπέρ. Το υπέρ των αριθμών του εισηγητή. Κατά, αποχές, εγκρίνεται το 670 με την τροποποίηση υιοθετείται, ε, λύνουμε και 33-32 της κυρίας Γκουλάρ. Την τροπολογία της Ίγκε, όχι, η Ίγκε πρέπει να ψηφιστεί. Η τροπολογία της Ίγκε πρέπει να ψηφιστεί, έχει δικαίωμα και όποτε ζητάει κάτι η Ίγκε το επιτυχάνει από τον πρόεδρο. Λοιπόν, 43-17 ε, σχόλια. Η συγκίτρια είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Υπάρχει μία πλειοψηφία υπέρ του 43-17 και συγχαίρουμε την Ίγκε. Περνάμε στην επόμενη σελίδα. σελίδα. 2.31. Τι είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επόμενη γραμμή 575. Είναι πολλαπλή τροπολογία ε, και οι δύο άλλες καλύπτονται. Το ίδιο ισχύει και για την επόμενη γραμμή. Production refunds for sugar used in the chemical industry. Περνάμε στο, στα άλλα μέτρα για το ελαιόλαδο 232 εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ του ελαιολάδου. Κατά. Ποιος προτιμάει δηλαδή βούτυρο. Αποχές. Εγκρίνεται 232. Περνάμε στο βαμβάκι. 233. Ποιος είναι υπέρ του βαμβακιού ποιος είναι ε, κατά οι γυμνιστές, ποιος ε, ε, απέχει. Το υιοθετούμε το βαμβάκι, άρα θα μείνουμε σοβαροί. Περνάμε στην εξαγωγή των φρούτων και ξαναέχουμε την 575 και Περνούμε στην επόμενη γραμμή, ε, η 4294 ελληνική, με τη στήριξη της εισηγητρίας. Υπέρ κατά, άποχες, εγκρίνεται. Και οι δύο οι επόμενες καλύπτονται. 4295, η ίδια ελληνική. Η εισηγήτρια είναι υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται και καλύπτει τις δύο επόμενες. School Fruit Scheme 220. Ε, Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Και καλύπτει και την επόμενη. Εδώ έχουμε πιλωτικά ε, σχέδια και πάμε στα export refunds for products of the wine growing sector. Το 575 είναι η πολλαπλή τροπολογία των πρασίνων. Γιατί λοιπόν να εξάγουμε ε, κρασί αν μπορούμε να το πιούμε. Περνάμε τώρα στην αποθήκευση του κρασιού. Storage of wine 41-76 η συγγήτρια είναι κατά. Εξαφανίζεται. Και αυτό λύνει το επόμενο. distillation of wine. Και πάλι έχουμε την πολλαπλή τροπολογία, άρα τίποτα δεν μπαίνει εδώ. Τώρα measure for alcohol το ίδιο. Aid for the use of must. για το μουστο δηλαδή. 41-79. Ο εισηγητής είναι κατά. Μήπως κάποιος είναι υπέρ του μουστου, όχι, άρα εξαφανίστηκαν οι μουστοι. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 80 ε, μάλλον στην επόμενη γραμμή γραμμή 41-80 του Γκόραν Φέρμ. Ποιος είναι υπέρ. Δεν τη στηρίζει ούτε ο κύριος Φέρμ. Ε, αρέσει στον Γένς, στην Γιούτα. Η Γιούτα είναι ανεξέλεγκτη τώρα. Αλλά δικαίωμά τη είναι ό,τι θέλει κάνει. Απορρίπτεται. Έχουμε μια συμβιβαστική. Μου λέγουν εδώ ότι στο 227 για το κρασί υπάρχει μια συμβιβαστική. Πράγματι, αυτό που πετύχαμε είναι να προσθέσουμε μόνο 10 εκατομμύρια ευρώ σε αυτή τη γραμμή. Μια προφορική τροποποίηση δική μου είναι στην τροπολογία 227 αντί 209 εκατομμύρια 300.000 να έχουμε 10 εκατομμύρια. Καταλάβατε όλοι. Θέλετε παρακαλώ να επαναλάβετε. Να καταψηφίσουμε την 227 και να, ψηφίσουμε, να ψηφίσουμε υπέρ της 496 ουσιαστικά. Donc, vous êtes en faveur Είσαστε δηλαδή υπέρ της 227, όχι, όχι. Είσαστε ε, υπέρ της 4296 και μας λέτε να ψηφίσουμε πρώτα τη 4296 και αν δεν υπερψηφιστεί θα δούμε. Ψηφίζουμε λοιπόν τη 4296. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεν μιλάμε πια για τις άλλες. Σε αυτή τη γραμμή είναι η μόνη πλειοψηφία η οποία υπερισχύει και καλύπτει τα πάντα. Ε, στο grabbing up scheme απορρίπτουμε μία τροπολογία χάρτων, στα other measures πάντοτε για το κρασί έχουμε μία τροπολογία 4181 του εισηγητή αλλά κανείς δεν το υπερασπίζεται και εξαφανίζεται. καλύπτει το 436 αλλά όχι το 235 το οποίο ψηφίζουμε ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και καλύπτει την επόμενη γυρίζουμε σελίδα 236 ο εισηγητής είναι υπέρ ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και καλύπτει την επόμενη 237 κατά αποχές εγκρίνεται και καλή την επόμενη. Dried fodder. Πρόκειται για ζωοτροφές, ξηρές ζωοτροφές, δεν ξέρω πώς λέγονται γερμανικά. Το 37 είναι χάρτον που διαγράφεται και το ίδιο ισχύει και για την πολλαπλή τροπολογία στο κάτω μέρος της σελίδας και περνάμε τώρα στο γάλα 579 τροπολογία πρασίνων που θεωρεί ότι υπάρχει υπερβολικό γάλα δεν είναι μία ε, πολύπλοκη τροπολογία αλλά ποιος είναι κατά αποχές απορρίπτεται και καλύπτει τις τρεις επόμενες που είναι ταυτόσιμες αλλά όχι τη 264 ο συγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ? Μοναχικός ο εισηγητής. Ποιος είναι κατά. Πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Το 264 η ηλεκτρονική ψηφοφορία μπορώ να ψηφίσω. Λίγη ψηφοφορία. Απερίφθη. Με 17 υπέρ 21 κατά. Η 262. Ο εισηγητής είναι κατά. Έχουμε όμως μία προφορική τροπολογία στο 262 εισηγήτρια. Έχω μία προφορική τροποποίηση για την παρέμβαση στα αποθέματα του αποβουτυρωμένου γάλακτος σαν συνέπεια των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα 10 εκατομμύρια να προτείνω στο αποθεματικό αντί 20 εκατομμύρια όπως προτείνει η Άγρη Επιτροπή Γεωργίας. Très bien. Donc on euh, oral pour Προφορική τροπολογία για να μειώσουμε ίστο στο ίμιση. Ποιος είναι υπέρ. Ηλεκτρονικά για την προφορική αυτή τροπολογία. Λίγη ψηφοφορία. Καταρρύπτεται και ε, υποβάλλουμε ε, την ε, πρόταση της Επιτροπής Γεωργίας. Κανείς δεν είναι υπέρ, άρα δεν θα το συζητήσουμε πλέον και περνάμε στο βούτυρο 218 ε, και εδώ έχετε προφορική τροπολογία Παρόμοια ιστορία προφορικά να τροποποιήσω το πόσο 25 εκατομμύρια αντί 50 εκατομμύρια ε, Cet amendement suscite la même majorité que tout à l'heure. Έχουμε την ίδια τις ε, ίδιες κατά σαν πριν, οπότε ε, καταρρύπτεται. 218, κάποιος υπέρ. Άρα δεν έχουμε ε, πλέον ούτε για την, ε, το γάλα σε σκόνη ούτε για το βούτυρο. Τώρα περνάμε στο γάλα στα σχολεία. School milk. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται και καλύπτει και την επόμενη day Fund το ο, περίφημο day Fund του Λάσλο Σόριαν ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας κατά ευχαριστώ έχουν τρελαθεί οι αντιπρόεδροι αλλά τέλος πάντων Οπότε η τροπολογία 219 εγκρίθηκε. «579. Θέλετε για τη 219 να γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση. Ωραία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία μπορώ να ψηφίσω εγώ. σταματήστε το. «25 υπέρ, 12 κατά». 579 είναι των πρασίνων. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Οι υπόλοιποι εκτός των πρασίνων. Απορρίπτεται. 238. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος άλλος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στο, στα βόδια και ε, στα μοσχάρια. Έχουμε την 575 που απορρίπτεται και τη 4184 του Γκόραν Φέρμ. Αλλά ο Γκέραν δεν το υποστηρίζει. Οι σοσιαλιστές είναι κατά πλην της Γιούτα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Άρα απορρίπτεται. Και καλύπτει την επόμενη και ψηφίζουμε την 239. Ποιος είναι υπέρ. Η συγκήτρια είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην επόμενη γραμμή. Έχουμε πάλι την πολλαπλή τροπολογία των πρασίνων που απορρίπτεται και θεωρούμε ότι καλύφθηκαν και όλα τα υπόλοιπα. Μετά, uh, refunds for pig meat. Για, δεν μας αρέσει το χοιρινό. Για τα αυγά δεν θέλουμε αυγά. Δεν μας μείνει τίποτα να τρώμε. Συνεχίζουμε τώρα. Πάμε στα πουλερικά. Δεν θέλουμε ούτε κοτόπουλο αλλά θέλουμε ε, τις ε, και, και το μέλι. Ποιος είναι υπέρ του 261 κατά εγκρίνεται 261. Τώρα έχουμε πιλωτικά. Άρα οι υπόλοιπες ε, δεν πρόκειται να εξεταστούν μέχρι την SPS. Η πρώτη είναι ε, Χάρτονγκ 4137 απορρίπτεται και μέχρι κάτω είναι οι κλασικές τροπολογίες Χάρτονγκ οπότε απορρίπτονται. Περνάμε στο Brief Special Premium. Τροπολογία 580 είναι για τις σταυρωματιχίες. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Για να ρωτήσω την εισηγήτρια. Η τροπολογία αυτή πολιτικά είναι υπέρ των ταυρομαχιών ή κατά. Να ξέρουμε δηλαδή. Οπότε η τροπολογία αυτή ο Τζέιμς. Πολιτική τροπολογία αυτή, πρόεδρε. Δεν θα μπορούσα να καθορίσω υπό όρους ε, προϋπολογισμού τι σημαίνει θανάσιμη έκβαση βρομαχίας; Δεν μπορώ να κρίνω το περί τίνος πρόκειται εδώ. James, να σε καλέσω σπίτι μου διότι στην περιοχή μου ή αν ο Σαλβαντόρ σε καλέσει στην Ισπανία ή πάσει προς το Γαλλία υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους διασκεδάζουμε με τους σταύρους οι μεν θανάσιμες οι άλλες όχι. Μπορεί λοιπόν ο καθένας να έχει τη γνώμη του. Είναι ένα πολύ λεπτό θέμα σε διορισμένες περιοχές. Άρα, ο εισηγητής, η ζητάει το λόγο όχι, είναι πλέον σαφές, μπορώ να το αναφέρω σε σχέση με τις παρατηρήσεις, αλλά είναι σαφές. Ωραία. Ποιος είναι υπέρ της 580, η συγκίτρια είναι υπέρ. Πρέπει να γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Θα ήθελα να ψηφίσω εάν κάποιος δεν θέλει να ψηφίζει από το ΕΛΚ. Λίγη ψηφοφορία. 18 υπέρ, 15 κατά και 7 αποχές. Οι 7 δεν είναι και πολύ θαραλέοι, λέει η κυρία Χάουγκ. Λοιπόν, πάμε στο, στην πρημοδότηση του καπνού. 620 συγγήτρια κατά ποιος είναι υπέρ. Ηλεκτρονική γιατί είναι οι σοσιαλιστές υπέρ, μπορώ να ψηφίσω εγώ προσωπικά. Ρωτάει ο πρόεδρος. 18 υπέρ, 20 κατά και 2 ο αποχές απορρίπτεται και καλύπτεται όλη η σελίδα εκτός από την 581 για τις πρωτεΐνες. Ποιος είναι υπέρ για το protein crops. Ποιος είναι κατά. Εγκρίνεται. Επόμενη σελίδα. 41-37 συνήθις χάρτονγκ. Τα ίδια. Το ίδιο και για το πρόγραμμα ΠΟΣΕΙ, αλλά πως, ε, ψηφίνουμε την τροπολογία Γκρελιέ 24 απορρίπτεται. 240, η συγκίτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 241. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 577 είναι ένα πιλωτικό. Ξεκινάμε από τη συνήθεια του κυρίου Χάρτον που απορρίπτεται. Η 200... 42. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται και καλύπτει και την επόμενη. 41-37 χάρτον θεωρείται καλυμμένη, 263 και 712 είναι πιλωτικά, θα τα δούμε αύριο και περνάμε τώρα στη 244. Ποιος είναι υπέρ. Κατά ηλεκτρονικά. Με συγχωρείτε. Από το όμως όμως αγχώθηκα. Και αυτό είναι η γραμμή Accounting Clearance of Previous Years. Θέλετε να ψηφιστεί τώρα κυρία ε, κυρία εισηγήτρια, δεν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε σαν παρέμβισμα, buffer line, άρα ψηφίζουμε την 544. Ε, Λίγη ψηφοφορία. 17 υπέρ, 22 κατά. Άρα εγώ δεν άλλαζα τίποτα και απορρίπτεται αυτή η τροπολογία και η επόμενη επίσης. Δεν έχουμε λοιπόν σε αυτή τη γραμμή τροπολογία και περνάμε στην επόμενη τώρα. Δηλαδή το πρώτο το οποίο θα ψηφίσουμε είναι το 245. Enhancing Public Awareness. Ποιος είναι υπέρ. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Ε, αποχές εγκρίνεται. στο τέλος ομάδος ε, δεν θα συζητήσουμε σήμερα ούτε για την αρχή της σελίδος 92. Ε, Μου είπαν ότι μέσω μίας τροπολογίας, μάλλον μίας συμβιβαστικής εχθές λύθηκε, όχι, με συγχωρείτε, 246, ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γυρίζω όμως σελίδα τώρα και πάω κατευθείαν στο Life Plus. Έχουμε τη συνήθη τροπολογία χάρτων που απορρίπτεται, αλλά έχουμε και την 431 που είναι μία τροπολογία για να διορθώσουμε τα σχόλια. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι δύο επόμενες καλύπτονται. Και πάμε στην 398, ε, ε, δηλαδή όλη η σελίδα μπορεί ε, να γυρίσει διότι πάμε, έχουμε είτε πιλωτικά είτε προκαταρκτικά. Το ίδιο ισχύει για την 94, για την 95. Πάμε στη σελίδα 96 κατευθείαν στην γραμμή Implementation of EU e Policy και Legislation on Climate Action. Ε, έχουμε μία συνήθη τροπολογία χάρτων, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε την 397. Είναι ο εισηγητής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και οι δύο επόμενες καλύπτονται η επόμενη σελίδα είναι πιλωτικά όλη η σελίδα 98 είναι πάλι πιλωτικά το ίδιο ισχύει και για τα 99 μέχρι τις αλίας, σελίες Φίσερις, Πρώτο μια τροπολογία Χάρτονγκ που θεωρούμε ότι απορρίπτεται αλλά πρέπει να ψηφίσουμε την 837 της Γκουε. Η συγγήτρα είναι κατά. Ναι, ναι, με συγχωρείτε, πάω πολύ γρήγορα. Λοιπόν, Λουίκ, έχει δίκιο, την 836 ε, Intervention in Fishery Product της Γκουε. Ποιος είναι υπέρ. Ορισμένοι είναι υπέρ οι φιλελεύθεροι. Αποχές απορρίπτεται λοιπόν. Το 837 της ίδιας ομάδος. Κάποιος είναι υπέρ. Όχι. Κανένας δεν είναι υπέρ. Απορρίπτεται. Γυρίζω σελίδα. Η 838 είναι πιλωτικό. Χάρτον απορρίπτεται. Όχι, όχι, είναι διαφορετική, συγγνώμη. Ασυνήθιστη τροπολογία, κύριε Γιάννησεν. Σε ποια σελίδα είμαστε. Είμαστε στην 100, αγγλικά. International Fisheries Agreements. Ο κύριος συνάδελφος. Συμφωνώ με τη μεσηλίδα 100, αλλά στη σελίδα 98 45, 46, 47 τις ψηφίσαμε. Κατά τη γνώμη μου δεν καλύπτονται. Καλύπτονται όλα. Τότε κάτι δεν πάει καλά με τον κατάλογο ψηφοφορία που έχουμε. Μου λένε ότι καλύπτονται οι τροπολογίε αυτέ. από τη συμβαστική στον Β1, στι γραμμε β Β1. Θα το ελέγξω και αν υπάρξει, ε, ε, ε, αν κάνω λάθος, θα το ψηφίσουμε αύριο. Λοιπόν, πού ήμασταν, ήμασταν στην 51. Επιτροπή ε, Αλίας. Η σύγητρα είναι υπέρ υπέρ. Κατά. Αποχές για την 51 εγκρίνεται. Συγγνώμη, συγγνώμη, πολύ συγγνώμη. Έπρεπε να ψηφίσουμε πριν την 51 και 41-46 χαρτών. Γιατί δεν είναι από τις συνήθεις τροπολογίες χαρτών. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52. Επιτροπή Αλίας. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 53 η υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σε 46 χάρτον όχι 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το πιλωτικό αύριο 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γυρίζω σελίδα. ...588... ...ψηφίζουμε... ...εισηγήτρια κατά... ...είναι κανείς υπέρ κανείς... ...α, συγγνώμη, είναι μερικοί... ...είναι Η πράσινη είναι υπέρ, είναι κανένα άλλο υπέρ. Και ο κύριο Χάρτον. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. 57. Επιτροπή Ελία. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 62. Η συγκεντρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η διάρρωση καλύπτουν της υπηρεσίας 63. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. ηλεκτρονικός έλεγχος για την 63. Κάνουμε φράγκα για κάτι το Σαλβαντόρα. Η Ούγγροι φυσικά είναι κατά της Αγγλίας. αταξίας στο ΕΛΚ. Οι φίλοι του ΕΛΚ ξέρουν τι θέλουν να κάνουν. Πέρας. 21 υπέρ 17 κατά εγκρίνεται. Όλη η επόμενη σελίδα θεωρούμε ότι καλύφθηκε. Το ίδιο και η πρώτη μισή σελίδα 104. 41 62 πρέπει. Ψηφίζουμε την 222. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε στην 2.23 Προφορική τροπολογία υπάρχει η συγκίδρια Είχαμε μια συμφωνία πρόσφατα σε σχέση με τις συζητήσεις του συντονιστής και αυτό, συντονιστές και αυτό είναι να δεχτούμε το αίτημα της Άγκρη για αυτό το κονδύλιο αλλά όχι 15 εκατομμυρίων το αίτημα αυτό το κονδύλιο αλλά 5 εκατομμυρίων διορθώστε με αν κάνω λάθος καταρχήν είναι η αποκατάσταση εδώ του προσχεδίου, να μην ξεπεράσουμε το προσχέδιο. Ευχαριστώ. Ο στόχος και αυτό που προτείνει η συγγήτρια είναι να αποκαταστήσουμε το σχέδιο του προπολογισμού. Αυτό θες συντόνια. Θες να επανέλθουμε στο προσχέδιο. Δεν είναι απόλυτα σαφές αυτό στο οποίο συμφωνήσαμε. Δεν είναι σαφές γιατί και για το αποθεματικό. Κάποιοι λένε κάτι και μετά ψηφίζουν διαφορετικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, αλλά εδώ πρέπει να είμαστε σαφέστατοι για το τι κάνουμε. Αν επανέλθουμε στο προσχέδιο προϋπολογισμού, αντί 15 εκατομμυρίων είναι συν 5. Αυτό νομίζω ότι ανταποκρίνεται σε αυτό που είχαμε συμφωνήσει. Αντί 15 είναι συν 5. Bien. Je crois qu'il y a un grand accord pour considérer que... Ακούσαμε τη σωστή ερμηνεία. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. Η γραμματεία κατάλαβε περί τίνο πρόκειται μάλιστα. Plant Health Measures, New Measures, 257 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οι δύο επόμενες καλύπτονται 258 εισηγείται υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τελειώσαμε με την κατηγορία 2. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά, αλλά είμαστε, έχουμε εξαντληθεί τελείως. Έχουμε μας χτύψει που μία. Δεν μπορούμε ουσιαστικά να ξεκινήσουμε με άλλο κεφάλαιο. Ραντεβού στις 3.

να προχωρήσω και μετά με αυτέ τι τρύπε που έχω δεν βγαίνει. Ήρμα Φίρστενμπεργκ δεν είναι αυτή η Δεν ε, θυμάμαι, αλλά στο σπίτι θα έχω είτε για τι μόδε αμερικάνικε είτε για τι αυτέ ε, ή για τα παρθούνε. Κάπου θα βρω σε κανένα περιοδικό και θα σου πω τα πόδια. Λοιπόν, τελειώσαμε το 2. Και εγώ δεν βγαίνω καθόλου από το κτίριο. Α, α, εγώ θα πάω στο σπίτι μου, το κλείνω ναι, μου.